So, äh, sehr geehrte Αξιότιμοι συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας και χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαστε τουλάχιστον δύο και έτσι μπορώ να σας μιλάω στον πληθυντικό, αγαπητοί συνάδελφοι. Χθες τα πράγματα ήταν ε, τραγικά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Πενταπλάσιο χρόνο χρειάστηκα για να καταφτάσω για τους γνωστούς λόγους, αλλά η σύνοδος του ΝΑΤΟ ευτυχώς από να τελειώνει. Ε, ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι για τον ε, προσκεκλημένο μας σήμερα το πρωί που είμαστε τόσο λίγοι και κλεκτοί ωστόσο. Να καλωσορίσω τον Βλάντισλαβ Γκορανόφ, εξ ονόματος της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας, της απερχόμενης. Καλώς ορίσατε. Και θα ήθελα... Σα ενημερώνουμε ότι επειδή για 37η μέρα 37 ημέρα συνεχίζουμε τις ε, κινητοποίησει μας κατά των ε, μονομερών συνθηκών εργασία που επιβλήθηκαν από τη δίκηση, θα παραχωρήσουμε προβάσεις ωραρίου σήμερα. Και να σα ενημερώσουμε, συνεχίζουμε τον Πρόεδρο, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά ζητήματα του τριμερίου διαλόγου, τα οποία εντοπίστηκαν χθε και όλο ιδιαίτερο η... το MRE και το θέμα των δευτερευόντων ΚΑΠ εντοπίστηκε ως ε, θέματα όπου οι απόψεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποκλίνουν ε, πολύ. Η επόμενη τριμερή διάλογη στις ε, 26 Οκτωβρίου και στις 6 Οκτωβρίου και έτσι δόθηκε σχετική εντόλη αυτά τα τεχνικά και θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε σήμερα το πρωί ως ε, συνήθως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε επί 10 λεπτά τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και μετά θα ακούσουμε επί 5 λεπτά έρωτα απαντήσεις με δυνατότητα επερωτήσεων εφόσον τηρείται το χρονικό όριο των τριών λεπτών. Στον πρώτο λοιπόν γύρο όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες οι πολιτικές ομάδες αυτές που εμφανίστηκαν εν πάση θα έχουν ε, τον προβλεπόμενο χρόνο τους και μετά θα ακολουθήσουμε το σύστημα don't. Αν μας μείνει χρόνο, θα συνεχίσουμε και με Catch the Eye. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον Βούλγαρο Υπουργό Βλάντισλαφ Γκορανόφ. Έχετε το λόγο. Ladies and gentlemen, the colleagues, uh, please prepare yourself. Κυρίες και κύριοι, προετοιμαστείτε να ακούσετε τα βουλγαρικά. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми членове на Комисията по економически... Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, πριν από έξι μήνες σας υπέβαλα και Σα παρουσίασα τι προτεραιότητε τη Βουλγαρική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών θεμάτων. Mm. Προηγουμένω, ε, είχα υπογραμμίσει και τον, ε, τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι ένα ε, σημαντικό παράγοντα για να πετύχουμε του στόχου μα. Σήμερα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα που επιτύχαμε από κοινού με όλες μα τι προσπάθειες ήταν σημαντικά για το απότερο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας δεν έγιναν ε, τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο για την αφοσίωσή σας και τον επικοδομητικό διάλογο ε, στις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Το κλίμα αυτό επικοδομητικής συνεργασίας πρέπει να συνεχιστεί για να έχουμε αποτελέσματα και στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Η Βουλγαρική Προεδρία με ανοιχτό πνεύμα και διαφάνεια έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να εξισορροπήσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Ακούσαμε και είχαμε πολλές διαβουλεύσεις με πυρογνώμονες ε, πολιτικό επίπεδο με τις ομάδες όλων των κατών μελών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα, οι ευρωπαϊκές επιποπτικές αρχές, οι ευρωπαϊκές ενώσεις ε, εταιριών και επιχειρήσεων, οι ενώσεις καταναλωτών, ε, μας ε, ε, βρήκαν και συζήτησαν μαζί μας 196 συναντήσεις. Το 15% όλων των συναντήσεων της βουλγαρικής προεδρίας. Τα θέματα εκοφήν ήταν 37 και στα 18 από αυτά καταλήξαμε σε κοινή θέση του Συμβουλίου σε κάποια πολιτική συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, οργανώσαμε, καταφέραμε μάλλον να έχουμε εξωσημείωτη πρόοδο στον τομέα τη τραπεζική νομοθεσία. Είναι ένα από του βασικού στόχου τη Βουλγαρική Προεδρία, όπω διατυπώθηκε στο κοινό πρόγραμμα του τρίου των Προεδριών, ήταν να επιτελέσουμε σοβαρή πρόοδο για να μειωθεί ο κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα με αντατικέ διαπραγματεύσει και πάνω από 200 πολυμερεί και διμερεί συναντήσει. Καταφέραμε να καταρτήσουμε μια κοινή προσέγγιση για το ε, πακέτο μέτρων ε, για τα τραπεζικά. Πετύχαμε συμφωνία σε περίπλοκα θέματα και εκεί όπου υπήρχε πόλωση σε σχέση με τις θέσεις των κρατών μελών. Ε, με την εισαγωγή κοινών κανόνων καταφέραμε να επιδιώξουμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εμπιστοσύνη για τον τραπεζικό τομέα. Ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε έτσι τις επιπτώσεις της προσφατότερης χρηματοοικονομικής κρίσης. Και Ελπίζουμε ότι θα έχουμε εντελεχέστερες και λεπτομερέστερες συζητήσεις για την κατανομή κινδύνου στο κεφάλαιο αυτό ε, προσεχώς. Τρεις μήνες μετά την ε, δημοσίευση της πρότασης κανονισμού για την αναθεώρηση του κανονισμού 924 και τα τέλη σε διασυνοριακές συναλλαγές ή την αντιστροφή των χρεώσεων, ε, είδαμε ε, να ε, εγκρίνεται η διαπραγματευτική εντολή από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι καλό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, διότι υπάρχει θέμα με τα τέλη των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρώ και με τι εθνικέ πληρωμέ σε νόμισμα των χωρών εκτός της Ευρωζώνης. Αξιοσημείωτη πρόοδος επίσης επετέχθη στο επίπεδο των για το σύστημα ε, προστασίας των καταθέσεων. Ε, στη διάρκεια διάφορων συναντήσεων είχαμε ε, θετικά αποτελέσματα και η Προεδρία πρότεινε μια εξισορροπημένη έκθεση πρόοδου για το θέμα αυτό. Στο νομοθετικό πακέτο για τα καλυπτόμενα ομόλογα, μόλις τα μέσα Μαΐου αρχίσαμε να εργαζόμαστε για το θέμα αυτό, δεν έχει επιτελεστεί πολύ πρόοδος αλλά συζητήσαμε το θέμα αυτό ε, λεπτομερώς και ετοιμάσαμε συμβαστικές προτάσεις για τον κανονισμό που αφορά την προληπτική μεταχείριση των ομολόγων και κάποια στοιχεία της σχετικής οδηγίας. Η Βουλγαρική Προεδρία ξεκίνησε τις εντατικέ διαπραγματεύσει σε δύο νομοθετικές προτάσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πρόοδος στον ε, τομέα αυτό έχει να κάνει και με την ε, επιδίωξη των προτεραιοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας για την μείωση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση μιας ε, αγοράς κεφαλαίων, μιας, αγοράς χρηματαγορών, μιας ένωσης χρηματαγορών και πρέπει να πω ότι η Βουλγαρική Προεδρία πέτυχε εξισορροπημένη πρόταση για την ε, νομοθετική νομοθετική πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό προϊόν. Ε, μετά τις συζητήσεις στο Κορεπέρ στις 19 Ιουνίου πήραμε διαπραγματευτική εντολή μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου και συζητήσαμε, θα συζητήσουμε με, τους, με τα συντεξιωτικά ταμεία και τους εκπροσώπους τους στο μέλλον στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Κυρίε και κύριοι, το Σεπτέμβριο θα ψεφίσετε για τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου επί του θέματο και ελπίζω ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί. Επίση, πετύχαμε στι συζητήσει ε, για τη δέσμη μέτρων για την άρνηση φραγμών στι διασυνοριακέ επενδύσει. Αυτή εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018. Μετά από εντατικέ διαπραγματεύσει πετύχαμε συμφωνία σε διαπραγματευτική εντολή με το Ευρωκοινοβούλιο η Βουλγαρική Προεδρία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Συστήματος ε, έδωσε μεγάλη προσοχή. Ε, πολλές συναντήσεις και ενδελεχής αναθεώρηση όλων των ε, παραμέτρων της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείναμε εναλλακτικές λύσεις και πετύχαμε σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις για την δεύτερη πρόταση που ε, επικαιροποιεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την υποδομή των ε, χρηματαγορών ε, την διάρθρωσή τους, κυρίως για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, την νομοθεσία ΕΜΗΡ οδηγία μας για ένα νέο μακροπροληπτικό καθεστώς για τους, επενδυτικούς, για τους επενδυτές διαμεσολαβητές ε, μεσάζοντες είναι κάτι που ε, επίσης προωθήσαμε και συνεχίζονται και οι συζητήσεις για τα τραπεζικά προϊόντα. Σε σχέση με την ε, πολιτική φορολογία είχαμε πολλές προσδοκίες και μεταξύ των πολιτών και συνεχίσαμε να δίνουμε έμφαση στα θέματα της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης και των επιθετικών φορολογικών συμφωνιών βάσει του οδικού χάρτη που ε, κατέρτισε η Προεδρία τον Ιανουάριο του 2018. Η Βουλγαρική Προεδρία ξεκίνησε να εργάζεται επί του θέματος με 7 ανοιχτά ντοσχέ όπου δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Η πολιτική συμφωνία το Μάρτιο του 2018 ε, προέκυψε στο επίπεδο της οδηγίας τάξη 6 που έχει να κάνει με τις διασυνοριακές ε, συμφωνίες. Αυτό από πολιτική σκοπιά ήταν πολύ σημαντικό, γιατί από τη μια επιδιώκεται περισσότερη φορολογική διαφάνεια, αποφυγή των επιθετικών φορολογικών συμφωνιών και εκφράσαμε την σταθερή μας ε, στήριξη προς την εφαρμογή κανόνων Το θέμα αυτό εξετάστηκε κατά προτεραιότητα και αναλάβαμε τη δέσμευση να πετύχουμε συμφωνίες στα δυνατόν συντομότερα. Συναντήθηκε τέσσερις φορές η ομάδα εργασία. και ε, επίση γι' αυτό συζήτησε και το Κορεπέρ. Πέντε από τα επτά κείμενα ε, αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας. Μετά από εντατική προετοιμασία, το ΕΚΟΦΗΝ πέτυχε συμφωνία για το κείμενο του συμβασμού και στις 25 Μαΐου Ε, το θέμα περατώθηκε. Σε σχέση με την φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, αυτό είχε εντοπιστεί ως προτεραιότητα της προεσδίας μας και 21 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή παρουσίασε μια δεσμή μέτρων για την ε, φορολογία της ψηφιακής οικονομίας το ε, αναλάβαμε το θέμα αυτό, οργανώσαμε συζητήσεις και το Μάρτιο σε άτυπο γεύμα του Κορεπέρ ε, προωθήθηκε μέχρι τον Απρίλιο που ανέλαβε η ομάδα υψηλού επίπεδου στις 18 Απριλίου. Στην άτυπη συνάντηση του ΕΚΟΦΕΝ στη Σόφια τον Απρίλιο 2018 το θέμα αυτό ξανασυζητήθηκε. πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή οικονομία ο φόρος για, τις ψηφιακές, για την ψηφιακή οικονομία και η συζήτηση ε, οργανώθηκε σε τέσσερις συναντήσεις λόγω των τεχνικών διατάξεων. Στις 13 Ιουνίου η ομάδα TAX υπέβαλε το πρώτο συμβαστικό κείμενο ε, για την πρόταση οδηγίας. Ως προς την κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείες υπάρχει ο χαρτής και βάσει των και έχει οριστεί η πορεία των εργασιών για το θέμα αυτό στην συνάντηση της ομάδας ψηλού επίπεδου τον Ιανουάριο του 2018. Η Βουλγαρική Προεδρία δήλωσε την πρόθεσή της να ε, πετύχει μια ε, εσωτερική φορολογική βάση όσο το δυνατόν πιο συνενετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω θα χρειαστεί και άρθρο προ άρθρο εξέταση του θέματο και μπορώ να δώσω και περισσότερε λεπτομέρειε αργότερα εφόσον χρειαστεί. Ω προ την έμεση φορολογία, έχουμε πετύχει το στόχο προτεραιότητά μα και εγκρίναμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέτρα αντιμετώπιση τη απάτης του φόρου προστιθέμενης αξία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό από πολιτική σκοπιά, διότι καταλαβαίνουμε ότι το να ενισχύσουμε την διοικητική συνεργασία θα περιορίσει τη φοροαπάτη. Ε, συμφωνήσαμε για τα ελάχιστα πρότυπα ε, του συντελεστή ΦΠΑ, 15% στα περισσότερα κράτη, ε, και κάναμε τεράστια προσπάθεια για να τελειοποιηθεί το ε, σύστημα που θέλουμε να προτείνουμε ως ε, τελικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακολουθήσαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλέπεται ειδικό καθεστώς για αυτές. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ήταν ένα ντοσχέ που επίση συζητήθηκε ω μέρο του πακέτου για το ΦΠΑ. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η συζήτηση ξεκίνησε στην αρχή τη Βουλγαρικής Προεδρία. Τη 9 Μαρτίου είχαμε διάσκεψη ψηλού επίπεδου στη Σόφια. Ανταλλαγή απόψεων ε, έλαβε χώρα εκεί. Τον Μάιο ξεκίνησαν οι τεχνικές εργασίε για το θέμα αυτό και η δική ομάδα εργασία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ανέλαβε τα ενία. Ε, η ομάδα εργασία θα λάβει την επόμενη εκδοχή του κειμένου στο Συμβούλιο και ε, τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω έχουν ήδη εντοπιστεί. Ε, όσο για τη σημασία των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων και για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίσαμε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων αυτών. Συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο κοινή προσέγγιση σχετικά και για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσαμε όπως προβλεπόταν ε, ε, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όπως λέγεται. Η ολοκλήρωση της Προεδρίας ε, δείχνει ότι τη δουλειά που κάνουμε την κάνουμε από κοινού. Δεν είναι ποτέ δουλειά ενός και μόνο κράτους μέλους. Είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας, ε, της δουλειάς μιας ομάδας συνεργατών και το σημαντικό είναι να ε, προέχει η θεώρηση που θέλουμε να έχουμε για το μέλλον, ε, μια θεώρηση μακροπρόθεσμη. Επίσης, ο πολιτικός διάλογος έχει σημασία, γιατί κάθε άποψη έχει τη βαρύτητά της, με την λογική ότι θα υπάρχει και υλοποίηση στην πράξη, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε, μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοράνο, για αυτή την ε, πολύ λεπτομερή αυτή εισαγωγή και να περάσουμε τώρα στις πολιτικές ομάδες. Από το ΕΛΚ, ο συντονιστής, ο κύριος Μπουρχαρτ Μπάλτ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχά να σα συγχαρώ και εσάς και την ομάδα σα και στι Βρεξέλλες και στην πατρίδα σα Ήταν πολύ επιτυχής η Προεδρία σα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Προεδρία σας ανέλαβε τα ενία της Προεδρίας σε μια εποχή κατεπίγουσας κατάσταση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό κανονισμό. Αναφέρατε ήδη ότι σε πολλά θέματα η Πρόεδρος Αλλά πολλά λοιπόν θέματα παραμένουν ακόμα ανοιχτά. Μία σύντομη λοιπόν ερώτηση από πλευρά σας, από πλευρά μας. Πού πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για ταχεία πρόοδο και ποιε ε, πιστεύετε ότι μπορούν να επιτευχθούν και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεδομένου του τελειώνει και η θητεία σε έναν χρόνο. Τι μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν στην τρέχουσα νομοθετική θητεία από πλευρά του Συμβουλίου Αυτέ είναι οι δύο ερωτήσει που είχα να σας απευθύνω και ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Θεωρώ ότι πολλά μπορούμε να πετύχουμε μέσα στη φοιτεία. και θα θέλαμε να το επαναλάβουμε. Θέλαμε να λύσουμε το γόρδιο δεσμό σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση στην Προεδρία μας. Το θέμα λοιπόν ήταν ε, αν θα στην μείωση του κινδύνου ή στην επιμερισμό του κινδύνου. Και σε αυτό δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Χάρη λοιπόν στις, ε, στη Γαλλία και στη Γερμανία ως βασικούς οικονομικής φορείς допълнителен напредък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 по отношение на корпоративната Σε ό,τι αφορά τώρα την εταιρική βάση προλόγησης, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για το ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μεγάλη πρόοδο, αλλά. Αλλά συζητήθηκαν διάφορες προοπτικές, διάφορες λύσεις και χρησιμοποιήθηκε μια συνέντευξη για να επιβληθούν κάποιες περιπτώσεις, κάποιες διατάξεις. Είχαμε κάποιους που μπλόκαραν κάποιες νομοθετικές αποφάσεις για να δείξουν ένα κράτος μέλος την αντίθεση του με ένα άλλο κράτος μέλος. Ελπίζω τέτοια φαινόμενα να μην τα δούμε σε πολλέ περιπτώσει και πολύ συχνά. Κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, ωστόσο, σημειώθηκε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, τα δημοσιονομικά, τους δημοσιονομικούς φακέλους. Πιστεύω ότι και ελπίζω η Αυστριακή Προεδρία να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Εργαστήκαμε σκληρά. Τα θέματα αυτά όμω είναι πάρα πολύ περίπλοκα σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικέ υπηρεσίε, σε ό,τι αφορά τι χρηματαγορέ. Και είμαι βεβαίως ότι μέσα στη θετία του Κοινοβουλίου αυτή θα σημειωθούν ε, επιτυχίες. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι στο τρέχον πουδουπού. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Μια και δεν έχει καταφτάσει ακόμα η κυρία Μπρέζ, δυστυχώ. Ε, θα πάρω το λόγο εγώ και λυπάμαι επειδή ασκώ και καθήκοντα προεδρία μία κάπω δυσάρεστη ερώτηση σήμερα το πρωί. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Βουλγαρική Προεδρία. Αφορά και την Αυστριακή Προεδρία, εξ όσων ακούσαμε, καθώ και τι επερχόμενε προεδρίε, σε ό,τι αφορά την Ειδική Διερευνητική Επιτροπή Τάξη 3, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και έτσι στο Κοινοβούλιο αυτό τα θέματα της φοροαποφυγή και όλων των νομοθετικών προτάσεων που συνδέονται με την φοροδιαφυγή θα εξεταστούν στην Επιτροπή αυτή, καθώς και τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της τάξη 1, τάξη 2 και της Επιτροπής για τα Panama Papers. Δεν θα είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ η οποία θα είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά. Δεν θα είναι η Καθήλυνα αρμόδια. Μάλιστα, η Επιτροπή Έκων, Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων δεν θα ασχοληθεί καθόλου με τα θέματα αυτά. Και αυτό θα πρέπει να το ορίσει το ίδιο το Κοινοβούλιο που θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργία του. Η Βουλγαρική λοιπόν Προεδρία κατά την ε, κατά το αίτημά μας να σας προσκαλέσουμε για να καταθέσετε στην Επιτροπή Τάξη 3 σε ό,τι αφορά και τα αποτελέσματα της Επιτροπής Πάναμα Τάξη 1 και Τάξη 2 και ποια θα είναι τα νομικά οι νομικές συνέπειες. Αρνήθηκε λοιπόν να έλθει στην Επιτροπή Τάξε γιατί δήλωσε ότι η αρμόδια είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποια επιτροπή είναι αρμόδια, για ποια θέματα και ε, δεν ε, τίθεται θέμα να το αμφισβητήσει αυτό κανεί εξωτερικό παράγοντά. Ε, το ερώτημα λοιπόν μου είναι κατά πόσον υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους η Βουλγαρική Προεδρία αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Επιτροπή Τάξη 3 και μία έκκληση προς τους εκπροσώπου τη Αυστριακή Προεδρία, προκειμένου να δεχτεί την πρόσκληση αυτή, την έκκληση αυτή. Γιατί πώ θα πείσουμε στην τελική ανάλυση τι ξένε διεθνεί εταιρείε να έλθουν να καταθέσουν στην Επιτροπή μας εάν το ίδιο το όργανο, το θεσμικό όργανο με το οποίο συνεργαζόμαστε δεν έχει αυτή τη διάθεση και αυτή την προθυμία να εισακούσει τις αιτήσει μας. Σα ευχαριστώ και καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώ. Όπω είπατε, στο Συμβούλιο αφιερώσαμε μεγάλο τμήμα των εργασιών μα και πολύ χρόνο στην φορολογία και, πολύ... και φαντάζομαι ότι και η Αστραϊκή Προεδρία θα συνεργαστεί ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Αλλά σε τελική ανάλυση έχετε δίκιο. Όταν λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει πώς, ε, ε, αποφασίζει πώς θα διοργανώσει τις εργασίες της και θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη εάν σας δόθηκε λάθος εντύπωση, αλλά το θέμα αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερως και εργαστήκαμε πολύ σκληρά από αυτό και πιστεύουμε ότι η ΕΚΟΝ είναι η επιτροπή στην οποία μπορεί να γίνει η συζήτηση αυτή. Ιδάλλως, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ενδεχομένως η Αυστριακή Προεδρία να έχει πιο πολύ χρόνο να ασχοληθεί και να δουλέψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ωστόσο, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ήθελα εγώ ως Υπουργός να αναλάβω την ευθύνη. Da δεν μας απασχολεί ποιος στέει. Μας απασχολεί να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία από εδώ και πέρα. Είναι παρανόηση αυτή που επικρατεί στο Συμβούλιο. Και θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να το διευκρινίσετε αυτό στο Συμβούλιο, ότι είναι μόνο δηλαδή η έκονα αρμόδια και η ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή, είναι αρμόδια για θέματα ξεπλήματο βρώμικου χρήματο, το οποίο συνδέεται προφανώ με τη φορά που πηγεί. Έχουμε και την νομική υπηρεσία, την Επιτροπή Γιούρη, η οποία ασχολείται ω καθήλυνα αρμόδια επιτροπή με πολλά νομικά ζητήματα σε διαφορά την ε, έκθεση αναχώρα. Έχουμε την Επιτροπή Κόντε, την Επιτροπή Ντέβε. Είναι διάφορε αυτέ οι επιτροπές για τα θέματα λοιπόν αυτά δημιουργήθηκε ακριβώς η τάξη 3, μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ακριβώς οι βουλευτές από όλες τις καθήλυνα αρμόδιες υπόλοιπες επιτροπές. Αν θα θέλετε λοιπόν να επιλύσετε αυτή την παρανόηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επόμενος θα ήταν ένας εκπρόσωπος του ECR, αλλά δεν βλέπω εδώ εκπρόσωπο του ECR, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ελεύθερους και στον κύριο Γέσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής Τάξε 3, Θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην, στις επαφές και συνομιλίες με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του και τους συναδέλφους του. Προσκαλώντας στην Επιτροπή Τάξε 3, εξήγησα ότι Ε, έπρεπε να δοθεί σημασία στον βασικό μας συνομιλητή. Το άκουσε και από τον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ, το άκουσε και από τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και ελπίζαμε ότι η Βουλγαρική Βουλή θα μπορούσε να ακούει ε, με την ε, δέουσα προσοχή του συνομιλητές της. Όπως είδατε, η Επιτροπή τα 6 συστάθηκε ε, επ' αυτού, διότι υπάρχουν απώλειες ενός 3 ευρώ από τη φορά που φύγει και φοραπάτη σε σχέση με τον ΦΠΑ. 75% των Ευρωπαίων θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη. Οπότε η τάξη 3 έχει μια σαφή εντολή ως Επιτροπή. Νομίζω ότι η Βουλγαρική Προεδρία από τη σκοπιά αυτή ήταν μια Προεδρία η οποία απλώς απέφευγε και υπονόμευε τη συνεργασία για το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου είναι, αφού αρνηθήκατε την πρόσκληση αυτή, την πρόσκληση την έλαβε η βουλγαρική κυβέρνηση, εσείς ο ίδιος στο Συμβούλιο και τώρα τουλάχιστον θα ε, διευκολύνεται την ε, συνεργασία με την ε, νέα Προεδρία, εξηγώντα την κατάσταση με έναν τρόπο κάπως πιο θετικό. Ναι, κι όμως αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο θέμα αυτό και νομίζω ότι έχει πάρει και διαστάσεις δράματος. Η απόφαση ήταν δική μου και είχε να κάνει με την δική μου κατανόηση του ρόλου αυτής της Επιτροπής ως Επιτροπής Εξεταστικής. Ανέκαθεν, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο με, για οποιοδήποτε θέμα, δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να αφιερώσουμε τώρα τόσο πολύ χρόνο ε, στο τι έγινε στο παρελθόν. Και αν με ρωτάτε ποιανού απόφαση ήταν όλα αυτά, ήταν δική μου η απόφαση. Έχεις άλλα λεπτά. Κοιτάξτε, κοιτάζοντας προς τα πίσω το τι έγινε με το θέμα, εγώ σας ερώτησα εάν θα διαμορφώνατε, θα μεταβάλλατε μάλλον τις τάσεις σας τώρα και τι θα γίνει με την Αυστριακή Προεδρία και τη συνεργασία για τα θέματα αυτά. Θα διευκολύνεται καθόλου. Κοιτάξτε, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, εγώ κοιτάζω προς το μέλλον. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τάξε 3 και επόμενος από τους πράσινους, ο κ. Ούρτασούν. Um, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θέλω να απηχήσω και εγώ τη φωνή της ομάδας μου και να τονίσω την σημασία της συνεργασίας με την Επιτροπή Τάξη 3. Σημαντικό είναι να κοιτάζουμε προς το μέλλον, αλλά αυτό θα το κάνει έτσι καλώς η Αυστριακή Προεδρία. Αλλαγέ θα επισυμβούν στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με τα φορολογικά, Υπουργέ. Η Προεδρία σας ήταν επιτυχής, πιστεύω ολοκλήρωσε την εξέταση του πακέτου για τη μείωση του κινδύνου. Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει το αν μας αρέσει το αποτέλεσμα ή όχι, αλλά ήταν μια επιτυχία. Για την φορολογία όμως τα πράγματα δεν προχωρούν με τόση ταχύτητα όσο θα θέλαμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω για τον φάκελο CBCR για την ε, αναχώρα υποβολή εκθέσεων. Και μας είπατε στην ε, εισηγήσή σας ότι εξετάστηκε αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι έγινε μόνο μια συνάντηση για το CBCR. Ε, θα θέλαμε να υπήρχε πρόοδος στο ντοσχέ αυτό. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες χώρες και ιδίως αυτές που αποτελούν τη μειονότητα που μπλοκάρει την πρόοδο του θέματος. Πιστεύετε ότι η επόμενη Προεδρία μπορεί να καταφέρει να το ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει η εξετασή του. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά κρατημέλη που έχουν ενδιασμούς και επιφυλάξεις. Θα το γνωρίζετε. Και δεν χρειάζεται να πω ποια είναι. Σε αυτή τη φάση, μια μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη για το ονομαζόμενο κείμενο που έχει παγώσει εντό εισαγωγικών, που έχει μπλοκαριστεί. Για το πώς θα προχωρήσουν όμως ζητήσεις του Συμβουλίου πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετά ανοιχτέ και διαφανείς. Ε, τα... Υπάρχουν κάποια κάτι μέλη που δεν θέλουν να απαρνηθούν τα πλεονεκτήματα που μέχρι τώρα και τα προνόμια που έχουν μέχρι τώρα τα φορολογικά τους συστήματα για να προφυλάξουν κάποιες εταιρείε και να συνεχίσουν να υποφελούνται από τα φορολογικά τους αυτά ε, προβαδίσματα. Δεν ε, ξέρω αν μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο επί του θέματος πραγματικά. Τουλάχιστον σύντομα. Εγώ τα συζήτησα επανελειμμένως ε, με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά πιστεύω ότι ακόμη και ο Αυστριακός Υπουργός, παρά την πολύ ε, μεγάλη του διάθεση να πετύχει πρόοδο, δεν είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρει κάτι. Έρνεστ. Ναι. Εφόσον έχουμε δύο λεπτά, να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση στον Υπουργό. Οι συζητήσει περί Ευρωζώνης. Είπατε ότι έχετε τη φιλοδοξία να προσχωρήσετε στο ευρώ. Ποια είναι η γνώμη σας μετά τις πρόσφατες δηλώσεις αυτά να προχωρήσουν τις επόμενους μήνες. Εμείς ε, αμφιβάλλουμε και ανησυχούμε. Και οι Ευρωπαίοι για την γαλλογερμανική πρόταση για τη λειτουργία της Ευρωζώνης και τον προπολογισμό ως ε, μελλοντικό μέλος ή μέλος που προσδοκεί να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη, η γνώμη σας θα ήταν πολύτιμη για το θέμα. Ναι, πιστεύω ότι μια στεναρή ευρωζώνη θα σημαίνει και μια ισχυρότερη Ευρώπη. Ως προς τη Βουλγαρία θα γνωρίζετε ότι βάσει και των συνθηκών έχουμε υποχρέωση να επιθυμούμε την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Πρέπει όμως να πληρούμε τις προϋποθέσεις Και υπάρχει και ένα σχετικό συμβούλιο για την νομισματική εξέλιξη στην Βουλγαρία ως προς την γαλλογερμανική πρόταση. Βρίσκω ότι σίγουρα δεν είναι άψογη, όμως δίνει, ε, δείχνει μια σωστή κατεύθυνση και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν την πρωτοβουλία να απαντήσουν ερωτήσεις και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επί σειρά ετών. Αυτά που αφορούν δηλαδή το μέλλον της νομισματικής ένωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είμαι βέβαιος ότι ο προπολογισμός εδώ θα είναι το βασικό ε, στοιχείο των μελλοντικών συζητήσεων δεν θα είναι και σημαντικότερη συνιστόσα που θα μείνει από τη γαλλογερμανική πρόταση. Συνολικά όμως πρέπει να πω ότι τις προτάσεις των δύο αυτών πρωταγωνιστικών κατών μελών τις υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ. Τώρα κανονικά θα είχαμε από την ΚΟΕ του Μιγγέλ Βιέγκας. Α, είναι εδώ. Έχεις το λόγο, Μιγγέλ. Καλημέρα σας. Έχω δύο ερωτήσει πολύ συγκεκριμένες η πρώτη έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος ή τα δημόσια χρέα, χρέη, που για πολλές χώρε χώρες αποτελούν ορολογιακή βόμβα, όπως για την Πορτογαλία παρόλο που έχουν αυξηθεί λίγο τα επιτόκια, εάν α, ε, ε, αλλάξει κάτι, μπορεί μια κατάσταση που τώρα μοιάζει ευνοϊκή, μπορεί να γυρίσει στο απολύτω αντίστροφο. Η Πορτογαλία είναι απλώ μια χώρα, δεν είναι μόνο που έχει αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη μα λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σα για το πώ προχώρησε το θέμα αυτό και το τι κινήσει έγιναν για την σταθερότητα τη Ευρωζώνη και την ειδικότερη κατάσταση τη κάθε χώρα. Πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πιο ειδική έχει να κάνει με το CCTV, δηλαδή έναν, ένα ντοσιά κλειδί που θα μπορούσε να επιλύσει πολλά ζητήματα σε σχέση με την εθνική κατάσταση και τη φοροδιαφυγή σε κάθε χώρα. Θεωρείτε ότι είναι ένα ντοσιά προτεραιότητας και ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και να βρεθεί κάτι ως λύση μέχρι το τέλος της δικής μας θητείας. Ναι, για τα δημόσια, για τα κρατικά χρέη. Είναι σαφώς πρόβλημα, Ιδίω για τις χώρες του Νότου. Η Βουλγαρία από τη δική της πλευρά είναι ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε 24% χρέος ως προς το ΑΕΠ και θέλουμε να το μειώσουμε σε 20% έως το 2020. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ε, γενιά που βρίσκεται στην αγορά εργασίας θα είναι έντιμη με τις επόμενες και θα ξοδεύει όσα κερδίζει και όχι παραπάνω. Ελπίζουμε λοιπόν οι χώρε σύντομα να φτάσουν σε κατάσταση να μπορούν να καλύπτουν το κρατικό του χρέο και να μην εξαρτώνται μόνο από την αλληλεγγύη. Βεβαίω, ω προ αυτό υπάρχουν προβλήματα και προκλήσει. Υπάρχουν κίνδυνοι και ρίσκα. Όμω, εάν γινόταν μια συζήτηση λεπτομερέστερη, Φαντάζομαι ότι η κατάσταση θα είναι πολύ ζωφερότερη από αυτά που σας λέγω τώρα. Ε, όμως, ε, για αυτό που έχετε εσείς κατά νου, αυτή την απειλή που διαφαίνεται, οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς. Ίσως πρέπει να είμαστε λιγότερο υποκριτές. Όταν κάποιος ε, παραβιάζει τους κανόνες και να μην είμαστε και τόσο ευέλικτοι όπως συχνά είμαστε. Παραείμαστε επί επίκης. Ως προς την κοινή εταιρική φορολογική βάση. Θα επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί. Τον Απρίλιο ξεκινήσαμε την εκπόνηση μελέτης αντικτύπου ε, για την κοινή φορολογική βάση. Καταρτήσαμε μια κοινή μεθοδολογία, μια κοινή υπόθεση εφετηρίας. Αυτή η μελέτη αντικτύπου προχωρά στις περισσότερες χώρες και έχουμε ορίσει μια βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ενδιαφερόμενες χώρες ε, για να ολοκληρωθεί και η μελέτη. Αυτό ήταν αρκετά απλό για την Βουλγαρία, γιατί έχουμε ένα πολύ απλό φορολογικό σύστημα. Ε, για την εταιρική φορολογία έχουμε χαμηλότερη βάση και γενικότερα. Η βάση μας είναι χαμηλή. Υποθέτω ότι οι πολιτικές σε κάποια κάτι μέλη θα επιζητούν κάτι, κάτι ανάλογο και προσπαθούν αυτό να το ε, πετύχουν μέσω μιας κοινή ευρωπαϊκής λύσης. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί τουλάχιστον σε αυτή, στη διάρκεια αυτής της θητείας. Διότι κάποια κρατημέλη εποφελούνται από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φορολογικού του συστήματος. Θα ε, αρπαχτούν λοιπόν από αυτά τα πλεονεκτήματα προσπαθώντας να τα κρατήσουν με χαμηλότερο συντελεστή στην ουσία. Αυτό επηρεάζει τι οικονομίε των υπόλοιπων κάτω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είμαι λοιπόν τόσο αισιόδοξο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να, να επιτελέσουμε ιδιαίτερη πρόοδο σε αυτό το θέμα εντό τη ε, θητεία. Ιδάλω, τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα κράτη και οικονομίε του θα επηρεαστούν Και είναι για κράτη που μέχρι τώρα τα φορολογικά του συστήματα έχουν φροντίσει να τα ε, οργανώσουν έτσι που να λειτουργούν καλά. Τώρα χρειάζεται κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Και μια και με τη διερμηνία υπάρχει μια μικρή χρονοκοθεστέρηση, είμαστε συνήθω 10 δευτερόλεπτα πίσω. Από το EFTD δεν έχουμε κανέναν, το ΕΝΕΦΕ, e από το ΕΛ και η e, ΕΒΑ Μαϊντέλ, αλλά δεν είναι εδώ. Ο Μπούρκαρτ Μπάλτ λοιπόν έχει πάλι το λόγο, συντονιστή. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στο ευρώ της χώρας σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πρόσφατα ότι η Βουλγαρία χωρίς αμφιβολία θα είναι η επόμενη χώρα η οποία θα προσχωρήσει στο ευρώ. Η χώρα σας τηρεί τα απαιτούμενα σε ό,τι αφορά τη σύγκληση στην παρούσα φάση και είναι έτοιμη λοιπόν να μπει στο ERM2 ακόμα και φέτος. Ωστόσο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατείνονται ότι η σειρά θα έπρεπε να είναι καταρχάς προσχώρηση στην Τραπεζική Ένωση και μετά να μπείτε στο θάλαμο αναμονής για να μπείτε στο ευρώ προσχωρώντας το ERM2. Αυτό προφανώς ε, έχει να κάνει και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται στα τελευταία χρόνια ο βουλγαρικός τραπεζικός ε, κλάδος ε, σε ό,τι αφορά την εμπορική τράπεζα κτλ. Η κρίση του χρέους, λοιπόν, μας έχει καταδείξει ότι όταν εκτιμούμε μία υποψήφια χώρα, αυτή η ευρεία εικόνα της οικονομίας είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, προκειμένου να αποφευχθούν αστάθειες κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Ερωτώ, λοιπόν, πού βρίσκεστε σε ό,τι αφορά το δρόμο προς το ευρώ ε, Πώς το εκτιμάτε και πώς εκτιμάτε και τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ε, σειρά των μέτρων. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι όντω το 2014 σημειώθηκε κρίση. Σημειώθηκε κρίση με μία από τι τράπεζε που αναφέρατε και με την Εμπορική Τράπεζα και υπήρξαν σχετικά επιχειρήματα γιατί τα stress test, οι δοκιμές αντοχής και η ποιότητα των αξιών δεν κατέδειξε κάτι το ανησυχητικό. Το 2016 έγινε επίσης και αξιολόγηση από την Παγκοσμία Τράπεζα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το συνολικό οικονομικό παγκόσμιο σύστημα και τα συμπεράσματα και τα πορίσματα της αξιολόγησης αυτής είναι δημόσια, ξέρετε, δεν εκτοδεικνύουν προβλήματα. Επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τώρα τις δηλώσεις των επιτρόπων, νομίζω ότι παρουσιάζουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητεί κανένα. Για παράδειγμα, ότι ε, σε κάποιο χρονικό διάστημα η Βουλγαρία θα προσχωρήσει στο ευρώ. Αν ε, μιλάμε μόνο για το χρονοδιάγραμμα, Υπάρχουν πρόκλησεις τα οποία οι νομοθετέ, θα πρέπει να κάτσουν να τα σκεφτούν για τη λειτουργία τη Τραπεζική Ένωση Δεν ε, έχει να κάνει με την ίδια τη συμφωνία που θα ρυθμίσει τη σειρά και τη διαδικασία ένταξης της χώρας στο ERM. Άρα δεν υπάρχει απαραίτητα σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής στην Τραπεζική Ένωση και τη, στην, στο ευρώ. Αυτό νομοθετικό πώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν ακολουθήσουμε το γράμμα και τον τύπο του νόμου, δεν υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση να βγούμε πρώτα στην Τραπεζική Ένωση πριν μπούμε στην ζώνη του ευρώ. Φυσικά και εκτιμούμε το γεγονό ότι Είναι αδύνατο να συμμετάσχει κανείς ε, στην Ευρωζώνη χωρίς να συμμετάσχει στην Τραπεζική Ένωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας νόμος ξεκάθαρος για τον ενοποιημένο εποπτικό μηχανισμό που να προκαθορίζει ότι αυτό αποτελεί την πρώτο βήμα για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη. Έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας, την τοποθετήσή μας και περιμένουμε από τους εταίρους μας ε, στην Ευρωζώνη να συμφωνήσουν με την τοποθέτησή μας για την ταυτόχρονη ένταξη στην Τραπεζική Ένωση και στο ERM. Φυσικά χρειάζεται και μια προπαρασκευαστική εργασία για να μπούμε στην Τραπεζική Ένωση. Αυτό εξαρτάται και από την ταχύτητα της όλης διαδικασίας. Μπορεί να πάρει έξι μήνες, μπορεί να πάρει 12 μήνες, αλλά εμείς θα ακολουθήσουμε με συνέπεια την πορεία αυτή με τη σαφή, ωστόσο, με το σαφή στόχο τη ένταξης στην Ευρωζώνη. Και ελπίζουμε να μην υπάρξουν ε, ε, μη νομιμοποιημένα επιχειρήματα όπως έγινε με τη ζώνη Σέγγεν σε ό,τι αφορά την ε, ζώνη του Σέγγεν γιατί αυτές οι αλλαγές ε, από οικονομικά σε πολιτικά επιχειρήματα, νομίζω ότι υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των βουλγαρών πολιτών στην λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση αυτή, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα από τον κατάλογο έχουμε και πάλι σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Η συντονίστρια, κύριε Μπερέση, είναι ακόμα στην κίνηση. Πολύ φοβούμαστε. Και θα ήθελα να την αντικαθιστήσω στην παρουσιαφάση, να κάνω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά το σύ... ΑΕΡ, το BRD, στην Προεδρία σας, όπως γνωρίζετε, το... ο φάκελος αυτός ολοκληρώθηκε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είμαι εγώ ο, ο εισηγητής για το CIR και το CDR και ο BRD είναι ο συνάδελφος ο κ. Φακμάρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, στις διαπραγματεύσεις προκύπτει ότι θα ε, υπάρχει μια δύσκολη σχέση μεταξύ της ε, χώρας υποδοχής και της χώρας ε, προέλευσης. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν θέλουμε να προβλεφθούν έγγραφα ρευστότητας. Εδώ που θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ τη ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση στο τελική ανάλυση αυτό διακυβεύεται και των λογικών αμφιβολιών των χωρών αυτών. Πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να συγκεράσουμε αυτά τα δύο σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά κεφαλαίου. Είναι διαφορετικές και οι απόψεις μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου Περιβάλλοντος έφτασε επιτέλους και ελπίζω να σε αντιπροσωπεύσα επάξια. Ε, είναι σαφές ότι η ερώτηση την οποία θέσατε είναι αρκετά ευαίσθητη. Είναι αρκετά δύσκολο, για να πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια συμβιβαστική λύση. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο για μένα να εξηγήσω σε ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο μπορεί η συμβιβαστική αυτή πρόταση να τροπολογηθεί και να αλλάξει μέσω της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω πάντως ότι η Αυστριακή Προεδρία θα τα καταφέρει και θα σημειώσει πρόοδο και στο συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα πάντως εδώ να τονίσω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια συμβιβαστική λύση και οι μελλοντικές συζητήσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας απευθύνω την έκκληση να δείξετε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Αλλιώς φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε και να ολοκληρώσουμε σύντομα. Σκοπός μας είναι να τα ολοκληρώσουμε αυτά στο δεύτερο ήμιση του έτους. Αυτό είναι σαφές. Ε. Και επίσης αυτό που είναι σαφές στην παρούσα φάση είναι να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έχω την εντύπωση ότι υπάρχει παρανόηση ότι έχουμε συναπόφαση Και όπως έχω διευκρινίσει επανειλημμένα, για κάθε αμετακίνητο σημείο ε, του Κοινοβουλίου έχουμε και του Συμβουλίου. Έχουμε λίγο χρόνο για το Catch the Eye. Έχουμε δύο λεπτά για τη δική σου ερώτηση και να δώσω το λόγο στο Catch the Eye. Θέλει κανένα να πάρει το λόγο. Να δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Well, I would like to congratulate the Bulgarian presidency ε, να ευχαριστήσω τη Βουλγαρική Προεδρία και τη Βουλγαρική Κυβέρνηση συγκεκριμένα. Γιατί νομίζω ότι τους ασκούμε κριτική άδικα για αυτά τα οποία συμβαίνουν με το φορολογικό του σύστημα. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ε, επιδείξει μεγαλύτερη εμπειρία και υπάρχουν άλλοι ισχυρότεροι παίκτες οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μάθω πώς η βουλγαρική κυβέρνηση επετυχαίνει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε ότι το ρωτάω αυτό γιατί προέρχομαι από την Ελλάδα. Έχετε ένα χρέος το οποίο δεν ξεπερνάει το 20 με 25% του ΑΕΠ. Εξαιρετικό. Έχετε επίσης πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα επιβολής φορολογίας, γύρω στο 10% ενώ στην Ελλάδα είναι 29% σχετικά με τα κέρδη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έχετε και θέματα με έλλειμμα. Ε, πώς θα καταφέρνετε λοιπόν. Πρόσωποι смислен при положение, че ние имаме 400 км. Κοιτάξτε, ευχαριστώ. Είναι ερώτηση ουσία. Είναι ερώτηση ουσία γιατί Εμεί έχουμε 1300 χιλιόμετρα α, ε, θαλάσσια σύνορα, Εσεί έχετε ούτε και εγώ ξέρω πόσα, ε, πολύ περισσότερα. Ίσως εδώ να έγκυται και η απάντηση. Τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο πιο οργανωμένα και πειθαρχημένα σε μας. Τώρα, στα πλαίσια των συζητήσεων στην Ευρωζώνη με τους εταίρους μας, μας λέγουν σύνεχως ότι συνορεύεται με την Ελλάδα, είστε γείτονες με την Ελλάδα. Λες και αυτό είναι αρνητικό. Εμείς είμαστε, όπως είπαμε, γείτονες, είμαστε πάρα πολύ κοντά η μία χώρα στην άλλη, αλλά δεν έχουμε εμείς σαν χώρα να ξοδέψουμε περισσότερα από όσα κερδίζαμε τα τελευταία χρόνια. Από πλευρά ορισμένων πολιτικών δυνάμεων η τάση αυτή στη δική σας χώρα κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα οι συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθούν, έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα, οδηγεί σε πάρα πολύ σκληρές καταστάσεις και οφείλεται να πληρώσετε το τίμημα για μια οικονομία λανθασμένη που ακολουθήθηκε και η οποία είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για τους πολίτες σας. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια πρόκληση σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής για την κυβέρνησή σας και για μένα είναι πρόβλημα και για τη δική μου κυβέρνηση είναι πρόβλημα, πόσο μάλλον για ε, την κυβέρνηση στην Ελλάδα πολλές φορές ε, και εμείς καμιά φορά αναβάλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και η αναβολή αυτή ε, θα μας οδηγήσει σε 10 χρόνια να τα αντιμετωπίσουμε μεγενθυμένα. Αλλά το θέμα δεν είναι να ασκούμε κριτική. Ε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική Ευρώπη θα πρέπει να σεβόμεθα τους κανόνες τους οποίους εμείς οι ίδιοι έχουμε αποφασίσει. Ας χρησιμοποιήσουμε το σεβασμό των αποφάσεων αυτών σαν μια σταθερή αξία και ας προσπαθήσουμε με ευφυΐα να μην ακολουθήσουμε κάποιες τάσεις οι οποίες ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, μας έδειξαν ότι αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο προπαρασκευασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο. η οικονομία σας ε, λοιπόν ε, με τα 13.000 χιλιόμετρα παραλίες που έχετε προφανώς κανένας ε, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι έχετε τη δυνατότητα να πάτε πολύ καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και κοιτάω και την ώρα και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κλείσω τη διαδικασία Καρσδιάη, να σας ευχαριστήσω κύριε Κορανόφα για την ε, παρουσίαση εδώ και για τις ε, ενδεχομένω δυσάρεστε ερωτήσει κάποιε φορέ ε, και εσά ενδεχομένω να μην μα ικανοποίησαν οι απαντήσει που ακούσαμε από πλευρά σα. Αλλά καλύτερα να ξέρουμε τουλάχιστον την αλήθεια και να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε και για την πρόοδο που πετύχαμε κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προ... και για την καλή συνεργασία με την Επιτροπή μας και ελπίζουμε να συνεχιστεί η ίδια τάση. Ευχαριστώ πολύ. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι λέω, να συνεχίσουμε στο 15 της ημερησίας διατάξης παρακαλώ. Στο 15 λοιπόν έχουμε τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2019, όλα τα τμήματα. Oh, ο συγκεκριτής μας είναι ο Ρούντεκ Νίντερμαϊερ. Γνωμοδότηση στην ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή BUDS ε, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας μηνύματα και θα ήθελα να δώσω το λόγο για 7 λεπτά στον συνάδελφό μας, τον Λούντεκ Νίντερμαϊερ. Λούντεκ, ευχαριστώ. Δεν θα χρειαστώ 7 ολόκληρα λεπτά Είχαμε ήδη μια συζήτηση, πρώτη συζήτηση νωρίτερα, υπήρξε και μια συνάντηση των σκιωδών με συμμετοχή αρκετών συναδέλφων και όπως τους υποσχέθηκα προσπαθώ να εντάξω ε, κάποιες από τις προτάσεις τους στο ε, δικό μας κείμενο. Τώρα έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος και σε επίπεδο κορεπέ Υπάρχουν κάποια κατεπήγοντα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα ας πούμε της ασφάλειας και της άμυνας. Οπότε εγώ δεν ζητώ υποχρεωτικά, αναγκαστικά περισσότερα χρήματα γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει περιορισμός εκεί αλλά μπορούμε να στοχεύσουμε στην αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των χρημάτων τα οποία είναι διαθέσιμα για την άμυνα, για την έρευνα στην άμυνα γιατί είναι σαφές ότι περισσότερες πιστώσεις δεν σημαίνει και καλύτερη ε, πρακτική εφαρμογή των πολιτικών μας. Εμείς και στα πλαίσια του διαλόγου με τα ΕΣΑΣ Προσπαθήσαμε και ξοδέψαμε αρκετά χρήματα για να καταλάβουμε τι είναι πίσω από τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και προσπαθούμε και στα πλαίσια της γραμμής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και οι αυξήσεις του προϋπολογισμού δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες σαν πρόταση. Μετά την εξέταση της κατάστασης και με τα ΕΣΑΣ και με το Συμβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι δημοσιονομικές συνέπειες θα έχει. Είπαμε λοιπόν ότι στο Κορεπέρ υπήρξαν προτάσεις να μειωθούν ε, κατά 100% κάποιες πιστώσεις για την EBA και την ΕΟΠΑ και 50% για την ΕΣΜΑ. Ε, νομίζω ότι σε σχέση με τα κάποιες από τις αποστολές των οργάνων αυτών, των αρχών αυτών, δεν θα ισχύουν λοιπόν του χρόνου και γι' αυτό ακριβώς μειώνουμε τις πιστώσεις σε κάποιες κατηγορίες κατά 50%. Και όπου χρειαστεί να διαφοροποιηθούμε θα το συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Όπως επίσης και 50% για προγράμματα στήριξης διαφορετικών πολιτικών. Εγώ εξεπλάγει γιατί από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και προτείνουν έτσι και αλλιώ ε, μια ουσιαστική μείωση των πόρων. Αλλά από ό,τι μάθαμε ε, για κάποια λόγω των προβλημάτων στην... της διεθνούς συγκυρίας γενικά επανερχόμαστε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν ε, την γραμμή αυτή. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία σε κάποιους τομείς προτείνονται μειώσεις κατά 23.000 ευρώ τι να σας πω τώρα, με εκπλήσει να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. Υπάρχουν και κάποια θέματα σε σχέση με την αύξηση της αποδοτικότητας κάποιων γενικών διευθύνσεων, δεν τα αμφισβητώ αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Όλα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου τις επόμενες ώρες, περιμένω όμως και τις απόψεις των κρατών μελών Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις προτάσεις τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι σχετικά δύσκολο γιατί θα πρέπει να κλείσουμε την τελευταία εβδομάδα του φθινοπόρου. Θα πρέπει να συνεργαστούμε κυρίως και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με mail Πάντως η συνεργασία ανάμεσα στους σκιώδεις μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ε, αν έχετε κάποια σημεία τα οποία θα θέλατε να συζητήσουμε, να με ενημερώσετε, αλλιώς ε, θα ψηφίσω, ασχοληθούμε με τις τροπολογίες μία προς μία. Ευχαριστώ το Λούντεκ για αυτή την επισκόπηση. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, στη θέση τη κυρία Μποναφέ, ο κύριος Χόνα Φερνάντες. Ναι, Πρόεδρε, όπως είπατε, δεν μπορεί να είναι εδώ η κυρία Μποναφέ και μου ζήτησε να την καταστήσω. Θα διαβάσω το σημείωμά τη. Πρόεδρε, συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησής του το κείμενο είναι σωστά εξισορροπημένο και ελπίζω να έχουμε θετικές συζητήσεις για να καταλήξουμε σε θέση της Επιτροπής. Όπως σημειώνει ο εισηγητής, πρέπει να τονίσουμε την ε, αξία του, ε, της χρηματοδότησης ε, που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ουσιώδης για τους πολίτες. Η άμυνα και ασφάλεια πολύ καλά ως προτεραιότητα από τον εισηγητή. Δεν θα έπρεπε όμω να είναι κορυφαία προτεραιότητα. Είμαι σοσιαλίστρια και δημοκράτη και από την ομάδα μα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην απασχόληση. Ε, δεν είναι απάντηση σε όλα ο νόμος των αγορών. Θα πρέπει να αναζητήσουμε βιωσιμότητα και κοινωνική συνοχή. Προσωπικός και με την έκθεση το πρωτοβουλία για, ε, για τα βιώσιμα δημοσιονομικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα ανάλογα νομοθετικά ντοσιά που έχουν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κατευθύνουν ε, την ε, οικονομική δραστηριότητα στην βιωσιμότητα. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα των πολιτών και το ανέφερα και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στην παρουσίαση των ε, διαφόρων προτάσεων της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τους επαρκείς πόρους για το συντονισμό και την παρακολούθηση των μακροοικονομικών ε, προτάσεων, θέλω να δοθεί έμφαση και στην ε, κοινωνική ε, διάσταση. Ένα βασικό στοιχείο του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η ομάδα μας θέλει αυτή η Ένωση να είναι πιο ε, αποτελεσματική στον αντίκτυπο που έχει στη ζωή των πολιτών. Για τις εποπτικές αρχές αναγνωρίζω τη θέση του εισηγητή για τον θετικό τους ρόλο και τη θετική του συμβολή, ιδίως για την ε, καλύτερη προστασία των χρηματαγορών και των καταναλωτών. Οι βασικές γραμμές πρέπει να επιτρέπουν ε, στους ε, αρμόδιους, αρμόδιες αρχές, με συντονισμένες προσπάθειες να καταλήγουν σε μια πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση. Σε μια κοινή εποπτική προσέγγιση ταυτόχρονα όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επιδιώκουν μια σωστή πρόθεση των ε, σκελών του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ακόμα και η χρηματοδότηση αυτών των αρχών, ακόμη και αν το δουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τη γενική αναθεώρηση, με απασχολεί μήπως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ μια παράγραφο για τη στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων ε, συμμετεχόντων στην αγορά. Όπως τονίζει ο στην έκθεσή του, Καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται το κόστος των υποπτικών ε, αρχών το 2019 γιατί έχουν αναλάβει και νέες αρμοδιότητες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αύξηση των κοντιλίων για τις εποπτικές αρχές, θα πρέπει οι σχετικές δημοσιονομικές γραμμές να αποφασιστούν αφού συζητήσουμε με τους αρμοδίους ε, προσώπους τους. Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλω ένα μικρό αριθμό τροπολογιών προκειμένου να ενισχυθεί και άλλο η γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε. Ε, ε, ευχαριστώ, Χώνας. Ευχαριστώ και για τα σχόλια τα οποία έκανες. και για την απουσία της κυρίας Μποναφέ. Η Κέιτ Σουίνμπερντ από το ECR είχε ζητήσει το λόγο, αλλά δεν είναι εδώ στην αίθουσα τώρα. Δεν φαίνεται όμως, οπότε δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής για τους φιλελευθέρους, για τους πρασίνους, ο Σβέν. Ούτε ο Σβέν ε, είναι παρόν στην παρούσα φάση και περνάω τώρα στην ΚΟΕ. Όχι, ούτε από την κούε κάποιος επιθυμεί να πάρει το λόγο. Συνεπώς λοιπόν φτάνουμε στο Catch the Eye. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους αν κάποιος από αυτούς θα ήθελε το λόγο. Κάποιος που δεν είναι στο κατάλογο των μελιδών, όχι. Μάλιστα. Να δώσω λοιπόν το λόγο πάλι στον Λούτεκ, στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Νομίζω ότι και άλλοι σκιώτε θα έρθουν σε επαφή μαζί μα για να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά τα σχόλια του συναδέλφου. Είχαμε πολύ περιορισμένο χώρο για την γνωμοδότησή μα. Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένες γραμμές, ε, σειρές που μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Αν θέλετε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ε, στις τροπολογίες, να δοκιμάσουμε να καταρτήσουμε και συμβαστικές τροπολογίες για να μην τα ψηφίσουμε όλα ένα προς ένα, γιατί νομίζω ότι οι τροπολογίες ε, επεκτείνουν την αρχική έκταση του κειμένου. Δυστυχώς είχαμε περιορισμούς. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κατά τα άλλα, να συνεργαστούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ελπίζω. Ευχαριστώ για το χρονοδιάγραμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προθεσμία για την κατάσταση για την γνωμοδότησή μας 18 ε, Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Και 29 Αυγούστου και 30 Αυγούστου θα κοιτάξουμε τις τροπολογίες. Ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, στις 29-30 Αυγούστου. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα μέχρι τις 10.30 μέχρι που θα καταστάσει ο Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς.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 Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Με τιμή και χαρά υποδέχομαι τον Ομοσπονδιακό Υπουργό, τον κύριο Όλαφ Σόλτς, σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να ανταλλάξετε απόψεις με τα μέλη της ΕΚΟΝ για αρκετά θέματα όπως και το πακέτο για την Νομισματική Ένωση και τα της Τραπεζικής Ένωσης και τους κρίσιμους φακέλους ε, με τους οποίους ασχολούμεθα σε αυτήν την αποφασιστική θα έλεγα φάση της ε, νομοθετικής μας εντολής. Η Ευρώπη έχει την δυνατότητα να κάνει κάποια θετικά βήματα έτσι ώστε να καταστήσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση ανθεκτικότερη, σταθερότερη και ικανότερη να βοηθήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή. Στις 19 Ιουνίου δημοσιεύθηκε η δήλωση προωθώντας ε, συγκεκριμένες θέσεις για μεταρρύθμιση της ε, νομισματικής ένωσης. Η δυνατότητα να μπορεί να απορροφά συμμετρικά σοκ ε, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε είναι κάτι με το οποίο έχουμε και εμείς συζητήσει, το οποίο έχουμε προτείνει στο παρελθόν. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως η ανάγκη να προωθήσουμε την διαδικασία μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο αλλά και την κατανομή και γενικά το διαμοιρασμό των κινδύνων όταν αυτό δημιουργεί θέματα σε κάποιους από μας. Γι' αυτό λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να σας μιλήσω για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν από κοινού. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα προχωρήσουμε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και κυρίως τις τράπεζες. Και εδώ έχουμε διάφορες βελτιώσεις οι οποίες ε, έγιναν τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες. Ε, αρκετή πρόοδος λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μαζέψει μια ορμή η οποία θα επιτρέψει κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν τόσο πιθανές τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη λοιπόν πρόταση που πετύχαμε θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη η οποία κατέστη δυνατή με το τραπεζικό πακέτο. Τα μέλη του ΕΚΟΦΗΝ συμφώνησαν επ' αυτού. Ξεκίνησε η διαδικασία τριμερών διαλόγων και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό αποτυπώνει μια καλύτερη ισορροπία αυτή που χρειάζεται για να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να υπάρχει και λιγότερο ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Το τραπεζικό πακέτο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αποτελεί μια σαφή συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό όλοι συμφώνησαν τελικά και πίστεψαν ότι πρόκειται για καλή λύση, την οποία μπορούσαν να υποστηρίξει, αλλά παράλληλα αποτελεί και την προϋπόθεση προκειμένου να καταστούν δυνατέ οι εξελίξει σε άλλου τομεί. Θα ήταν μεγάλη παρανόηση να θεωρήσουμε ότι το τραπεζικό πακέτο με τα διάφορα κριτήρια τα οποία αναφέρονται δεν θα υλοποιηθεί. Και αν δεν υλοποιηθεί, θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τις άλλες δυνατότητες που συζητάμε σήμερα, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τα υπόλοιπα. Αν δεν γίνει το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά την ποιότητα ενός ανταγωνιστικού, παγκόσμια ανταγωνιστικού τραπεζικού μοντέλου, θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα. Και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερως στις διάφορες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την ε, ανάγκη να, υπάρχει, να υπάρχουν διαθέσιμα ποσά τα οποία να χρησιμοποιούν σε περίπτωση κρίσης. Αν μειωθούν λοιπόν αυτές οι απαιτήσει, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ μακριά ατζέντα η οποία δεν θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι το τραπεζικό πακέτο το οποίο αποτέλεσε καρπό διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και το οποίο υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι θα ήταν η πιο σημαντική συμβολή στην ολοκληρώση της ε, τραπεζικής αυτής Ένωση την οποία χρειαζόμαστε. Κατά τα άλλα είναι σωστό αυτό που είπατε. Χρειαζόμαστε περαιτέρω πρόοδο για να αναπτυχθεί αυτό το τραπεζικό πακέτο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς ε, θα συμφωνήσουμε για την μεταξέλιξη του μηχανισμού σταθερότητα του ESM. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε και να τονίσω ποια είναι τα πιο σημαντικά. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές Καλό είναι να γίνουν σε ένα βήμα, γιατί άμα αλλάζουν τα πράγματα διαρκώς 5-6 φορές, δεν θα υπάρχει καλός αντίκτυπος. Να τα μαζέψουμε όλα αυτά λοιπόν, να τα συζητήσουμε και να τα επιβάλλουμε με μιας. Να υπάρξει τροποποίηση και της συνθήκης, η οποία να προετοιμαστεί και σωστά Και γι' αυτό λοιπόν αναπτύξαμε και μια πρόταση με τον Γάλλο συνάδελφο και την οποία και συζητήσαμε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το πρώτο λοιπόν ε, σημείο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντα ε, ενό Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό, γιατί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση των χωρών που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην πρόσβαση στι ε, ε, αγορέ και η Ελλάδα ολοκληρώνει το πρόγραμμά της ε, είναι μεγάλη ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν αποτελεί ένα μικρό περιφερειακό πρόγραμμα ε, στην Ευρώπη. Όχι, ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο ε, σταθεροποιεί την Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι είναι σωστό να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό και να δώσουμε τέτοιες δυνατότητες περαιτέρω. Χρειαζόμαστε να λεφτούν αποφάσεις ότι αφορά τη μεταξέλιξη της τραπεζικής ε, δομής. Έχουμε τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και ότι αυτό συνεπάγεται για την εξασφάλιση των τραπεζών. Αυτό το συζητάμε εδώ και καιρό. Χρειαζόμαστε μια σταθεροποίηση προκειμένου να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη σταθεροποίηση των τραπεζών. Αυτό το σύστημα ασφαλείας, το κοινό backstop, θα πρέπει να κατοχυρωθεί μαζί με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Άρα, αν ε, μεταξελιχθεί αυτή η λειτουργία ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητα και του Μηχανισμού Ασφαλεία, θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την απαραίτητη μεταρρύθμιση. Και αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην παρούσα φάση είναι το εξή. Να απελευθερώσουμε τον μηχανισμό σταθερότητα από μια λειτουργία που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, από την άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί αυτό νομίζω ότι θα απελευθερώσει το μηχανισμό, γιατί θα απελευθερώσει πόρους που ε, φυλάσσονται για, για ένα σκοπό που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Και το ίδιο ισχύει και για το θέμα του τι κάνουμε σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα. Πιστεύουμε ότι εδώ χρειαζόμαστε ένα κοινό καθεστώς για να πούμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα α, να γίνει συνολική αναδιάρθρωση του εθνικού χρέους και να υπάρξει μια αναδιοργάνωση. Αυτό είναι δυνατόν λοιπόν. Και αυτό θα συνέβαλε στην ε, περαιτέρω σταθεροποίηση του συστήματος. Τι άλλο περιλαμβάνεται προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τι θα γίνει στο μέλλον με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό θα πρέπει να το εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν. Ε, υπάρχει λοιπόν ανάγκη να συζητήσουμε ποια είναι η στοχοθεσία, ποιοι είναι οι στόχοι. Σε ό,τι αφορά το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μιλάμε για 5% σε μεικτό επίπεδο και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τι έχει συμβεί σε ιστορικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε διαφορέ χώρε πώ έχουν εξελιχθεί και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε αξιόπιστε συμφωνίε, μεμονωμένε, οι οποίε στη τελική ανάλυση θα μα οδηγήσουν σε μια κοινή διαχείριση τη κατάσταση στι ε, τράπεζε που πλήττονται από το θέμα αυτό. Και αυτό πιστεύω ότι θα ήταν μια ευλογή ανάγκη. Όλα αυτά λοιπόν από κοινού πιστεύω ότι θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε γρηγορότερη υλοποίηση του συστήματος ε, ε, του μηχανισμού ασφάλειας του backstop πριν από το 2024 και νομίζω ότι σωστό θα ήταν να ισχύσει αυτό για όλους ταυτόχρονα. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των μεμονωμένων χωρών και των μεμονωμένων τραπεζών. Δεν θα ήταν θετικό να συμμετέχουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι όχι. Να γίνουν όλα λοιπόν ταυτόχρονα σε ένα βήμα. Αυτό είναι άλλωστε και η πρότασή μας και άλλα θέματα παίζουν κάποιο ρόλο. Το έντις, για παράδειγμα, όπου σίγουρα θα πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Θεωρούμε ότι καταρχάς θα πρέπει να συζητήσουμε τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη και φυσικά πολλά θέματα συνδέονται με το έντις, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που χρειαζόμαστε, πιστεύω. Και πρέπει να σκεφτούμε επίσης ε, τις δημοσιονομικές ικανότητες, πώς θα λάβουν χώρα. Έχουμε διάφορες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Πολλές είναι ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέρουσες. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει και με τους Γάλλους ομολόγους, τους Γάλλους φίλους μας και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα και απαραίτητα εργαλεία. Αυτά που είναι σαφή για μας, να σας τα αναφέρω στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κινηθούμε. Να μην ε, συζητήσουμε δηλαδή ε, συστήματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά αυτά ζητήματα. Επίσης σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαμόρφωση λοιπόν των προτάσεων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιες προτάσεις ένα από τα στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε είναι κατά πόσον θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια αντασφάλιση στα πλαίσια της ε, ασφάλισης ανεργίας. Αυτό θα έχει και λειτουργία σταθεροποίησης σε δύσκολους ε, καιρούς. Αυτό είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα, γιατί σε τελική ανάλυση είναι το σύστημα το οποίο εφαρμόσουν οι ΙΠΑ για την ασφάλεια ανεργίας. Και Υπάρχουν και κάποιοι όροι που συνδέονται με το σύστημα αυτό. Τα κράτη λοιπόν θα πρέπει να έχουν συστήματα προστασίας των ανέργων, αλλά σε περιπτώσεις μακροοικονομικών κλειδονισμών ξεσπάσματος μιας ξαφνικής κρίσης, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να παρέχει αλληλοβοήθεια και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το συζητήσουμε πιο επισταμένο, Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι στην παρούσα φάση μπορεί να επιτευχθούν μεγάλοι πρόοδοι, μεγάλες εξέλιξεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά που έχουμε να συζητήσουμε άμεσα, το τριμερή διάλογο για το τραπεζικό πακέτο που θεωρώ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, επί της βάσης των όσων συμφώνησαν τα ευρωπαϊκά κράτη, να κάνουμε τις περαιτέρω τα περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθεροποίηση ε, και παράλληλα να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης ε, στα πλαίσια των δημοσιονομικών ικανοτήτων. Αν λοιπόν τα αναπτύξουμε όλα αυτά, πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα που ήταν πολύ ωφέλιμο. Και όπως είπα εισαγωγικά, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Έχουμε μια νέα ορμή έχουμε αποκτήσει μια κεκτημένη ταχύτητα στην Ευρώπη και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να περάσουν μέτρα τα οποία θα είναι χρήσιμα. Έχουμε επίσης ε, καλά οικονομικά στοιχεία, το ξέρατε όλοι ότι πολλές χώρες ε, εκπληρώνουν τα κοινά κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει. Είναι λοιπόν η χρονική στιγμή που πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω το πρόγραμμα, το σύστημα προκειμένου να μπορούμε να αντιδρούμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την πληρέστατη παρουσίασή σας και την παρουσίαση περίπτωση, των γερμανικών θέσεων. Ήταν ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Ε, εμείς ως ε, εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση γίνεται με βάση δύο κείμενα ισότιμα και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις ένας ε, τριγωνικός διάλογος δεν είναι ποτέ ή όλα ή τίποτα. του, η πίεση ε, μαζική του ενός οργάνου εις βάρος του, άλλου. απλά πρέπει από κοινού να εντοπίσουμε τα στοιχεία στα οποία μπορεί να υπάρξουν συμβιβαστικές προτάσεις. Έτσι δουλεύουμε σε επίπεδο νομοθετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία αναφερθήκατε που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οι συνάδελφοι είναι σαφές ότι θα τα σχολιάσουν. Μπάλτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βρίσκεστε σήμερα στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων και εγώ προσωπικά χαίρομαι που είναι εδώ ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών στην τελευταία μου συνεδρίαση ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρέπονο. Ο κύριος Λάγκε λέει διάφορα εκτός μικροφώνου. Αστείευεται ο κύριος Μπάλτς. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η επισκόπηση που μας δώσατε. Να σας ευχαριστήσω για αυτήν. Και να πω ευθύ εξ αρχής ότι συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμησή σας ότι τώρα έχουμε την ε, απαραίτητη ταχύτητα, διεκτημένη ταχύτητα, την οποία και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Εκ παραλλήλου, γνωρίζω παράλληλα πόσο ευρείες είναι οι αξιώσεις και οι προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και εγώ από δική μου πλευρά να πω το εξή. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ESM και του backstop του μηχανισμού του συστήματος ασφαλείας. Τι πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον είναι ρεαλιστικά υλοποιήσιμο, τι μπορούμε να πετύχουμε, γιατί φυσικά πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ορμή. Το 2019, για παράδειγμα, με τις ευρωεκλογέ, τη νέα σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, εκ νέου ανάληψη λειτουργιών ε, κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε διάφορα στοιχεία. Άρα, πού πιστεύετε ότι βραχυπρόθεσμα, πέρα και από αυτά που διευκρινίσατε, μπορούμε να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πρόοδο. Κάτι άλλο που έχω να ρωτήσω, η συνάδελφο Περβάνου Περέ και εγώ του τελευταίου μήνε εργαστήκαμε για τι νέε ε, εκθέσεις για τις νέες αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, των ESAs. Ερωτώ λοιπόν από πλευρά του Συμβουλίου ως Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, πιστεύετε ότι υπάρχει απαραίτητη βούληση και προθυμία στους κόλπους του Συμβουλίου για να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο και να καταλήξετε μέσα στην τρέχουσα θητεία σε κάποιες συμφωνίες, γιατί δυστυχώς έως τώρα από πλευρά του Συμβουλίου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δισταγμοί καθυστερήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα μα ενδιαφέρει να ακούσουμε ποια είναι η άποψη του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Αυτό που προσπάθησα να σας παρουσιάσω ήταν ε, ε, μια πληθώρα ζητημάτων, μεγάλη και ευρεία ατζέντα. Νομίζω ότι η φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να συμφωνήσουμε ό,τι εντάσσεται στο τραπεζικό πακέτο και με το μηχανισμό σταθερότητας και όλα όσα συνδέονται με αυτόν για τις άλλες δύο συζητήσεις. Θα πρέπει και εκεί να προχωρήσουμε γρήγορα, αλλά ενδεχομένως να μας πάρουν πιο πολύ χρόνο, γιατί θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία συνένεση για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα μέτρα και είναι διαφορετικέ οι απόψει των κρατών μελών, διαφορετική και η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήταν καλή πρόοδος αν θα συζητούσαμε την δημοσιοοικονομική ικανότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς θα ταιριάξουν μεταξύ τους και πώς θα διαμορφωθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ πιστεύω ότι αυτό που είναι σημαντικό για πολλούς εξημών είναι τα εργαλεία τα οποία θα σχεδιαστούν να μπορούν να αντιδρούν σε συγκεκριμένες ε, καταστάσεις. Ε. Αλλά παράλληλα να δημιουργηθεί και ένα καθεστώς, μια κατάσταση στην οποία θα έχει κάθε χώρα και την δική της ευθύνη για τη μοίρα, τη της. Και όσοι είναι διστακτικοί σε ό,τι αφορά αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα, πιστεύω ότι αν γίνει σωστά ο σχεδιασμός ε, θα περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία γιατί θα αυξάνει τη σταθεροποίηση και τη σταθερότητα των, ε, α, της κατάστασης χωρίς να άρει την ευθύνη της κάθε χώρας. Αυτό που θα παίξει ρόλο στην όλη συζήτηση είναι η σκέψη του κατά πόσον ε, σε ό,τι αφορά και τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Το συζητάμε αυτό εκ νέου μεταξύ των κρατών μελών. Και νομίζω ότι δύο περιστατικά βοηθούν την όλη συζήτηση. Το ένα το λέω ξεκάθαρα, είναι η χειρονομία του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος είπε ότι το φορολογικό μοντέλο το οποίο ακολουθεί η Γαλλία, αν το ακολουθήσουμε, και αν συμφωνήσουμε να χρησιμοποιηθεί για ευρωπαϊκούς σκοπούς και ανέφερε διάφορους, σε διάφορες περιστάσεις, αλλά και η συζήτηση για το κατά πόσον αυτό μπορεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν καθιστά τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα, γιατί ξαφνικά έχουμε μία προοπτική. Τα κράτη μέλη να έχουν κάτι από τις ε, συμβολές των κρατών μελών. Η Γερμανία λοιπόν θα ε, μείωνε την εισφορά της και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει καταλήτη για να πετύχουμε μια συνένεση. Πιστεύω λοιπόν ότι η σύνδεση της πρότασης αυτής με το γεγονό ότι πρέπει να συζητήσουμε και θέματα προϋπολογισμού ίσως να δημιουργείται συνθήκες για να πετύχουμε την πρόοδο αυτή. Επίσης κάτι άλλο που συζητήσαμε θα θέλαμε και στο θέμα να, να σημειωθεί πρόοδο και σε ό,τι αφορά και τον κοινό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό, το θέμα των υποπτικών αρχών. Εδώ χρειαζόμαστε πρόοδο, να δούμε τι θα πετύχουμε, τι μπορούμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των εθνικών καθεστώτων και των ευρωπαϊκών αρχών για να μην δημιουργήσουμε νέα γραφειοκρατία νέες ε, ανεπάρκειες. Ε, αλλά από ό,τι είδα έχετε επικρίνει και κάποιες από τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Περές και θα σας ζητούσα να τηρήσετε το χρονικό όριο των δύο λεπτών. Με προσκαλείτε να πάθω φρούστρα εξ αρχής. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Πρέπει να διαλέξω. Θα σας ρωτήσω για το τελευταίο που είπατε. Τη δημοσιονομική δυνατότητα. Και αναφέρατε και τις ε, πρόσφατες δηλώσεις όπου υπάρχουν και κάποιες διαβεβαιώσεις για την ε, ανεργία Πώς θα εργαστείτε για να εμβαθύνετε αυτές τις προτάσεις και να ενταχθούν στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωζώνης, αλλά και για το όσα συζητάμε τώρα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ένα τοπίο όπου δεν θυμόμαστε αρκετά ότι η βαρύτητα της Ευρωζώνης, το ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Brexit θα περάσει από το 73 στο 86%. Κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τι επιτακτικέ ανάγκες που θα πρέπει να ικανοποιεί η Ευρωζώνη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτέ τι διπλωματεύσεις επειδή μιλήσατε και για το κοινωτικό επίπεδο. Και επίση, αυτή η πρόταση πώ θα διαρθρωθεί με αυτή που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν μηχανισμό στήριξη των επενδύσεων ε, στο σκέλο τη σταθεροποίηση. Διότι ξέρουμε ότι το ένα δεν μπορεί να μην συμβαδίζει με το άλλο. Ποια είναι η πρότασή σα λοιπόν για να προχωρήσουν παράλληλα αυτά τα δύο. Πώ θα στηρίξουμε τι επενδύσει για να μπορέσουμε εν τέλει να καταλήξουμε στη φιλοδοξότερη και απαραίτητη ε, αυτή ε, πρόβλεψη για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την ανεργία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ερωτήσει αυτέ και να προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. καταρχά θα πρέπει να συζητήσουμε και το σύστημα, το, το σκοπός ε, της ε, αντασφάλισης αυτής ε, για τις ανέργους και καταρχάς να μιλήσουμε ότι δεν διευκρινίσουν δεν πρόκειται για ένα σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των ανέργων. Αυτό θα ήταν όνειρο απατηλό πιστεύω. Αλλά να υπάρχει μία ασφάλιση λοιπόν σε ό,τι αφορά το κόστος ε, χρηματοδότησης της ανεργίας για να μπορεί να αντέξει ας πούμε, μια χώρα για δύο χρόνια. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός αυτός. είναι ανοιχτό ακόμα αυτό στις προτάσεις, ε, αλλά το γεγονός ότι το συζητάμε καν αποτελεί μεγάλη πρόοδο. Το πώς ε, σχετίζεται αυτό με το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα αυτόνομο σύστημα, ανεξάρτητο σύστημα, το οποίο δεν παίζει απαραίτητα ρόλο, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών ικανοτήτων ενδεχομένω. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω αυτό που είπατε. Το θέμα του ποια θα είναι στο μέλλον η σημασία του ευρώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το εκτιμήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει μια συνέπεια αυτό που αναφέρεται για το 85% το οποίο θα δημιουργείται στην ε, Ευρωζώνη. Θα είναι όλο και μεγαλύτερη η ελκυστικότητα της Ευρωζώνης και αυτό θα οδηγήσει σε νέες συζητήσει οι οποίες ε, δεν μπορούμε φυσικά να τις προβλέψουμε στην παρούσα φάση, αλλά θα πάρουν το δρόμο τους σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Είναι ενδιαφέρον γιατί θίγει το θέμα του κατά πόσον το συγκεκριμένο αυτό μοντέλο είναι το πλέον κατάλληλο. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και καλό θα είναι σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει επικάλυψη με τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι έχει νόημα να γίνεται, τι γίνεται με τις πιστώσεις ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά τα παιδεία, τα θεματικά παιδεία αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε πιο επισταμένως και να δούμε τι θα προκύψει μετά από την ενδελεχή αυτή εξέταση. Thank you, Joachim Ευχαριστούμε κύριο Σταρμπάτη. Κύριε Υπουργέ, καταρχά να σα ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ για να μα απαντήσετε. Πριν από ένα χρόνο, ο τότε Ιταλό Υπουργό Οικονομικών στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων μα παρουσίασε το όραμά του για την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης ε, Ανέργων και μας είπε ότι σε περίπτωση προβλημάτων ε, ισοτιμίας ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή ασφάλιση για την ανεργία. Και τότε λοιπόν θέλετε τώρα μάλλον να ε, μην συμπεριληφθεί η διατύπωση ανακατανομή. Και μιλάτε λοιπόν για μια τέτοια αντασφάλιση. Αυτό τι σημαίνει ότι οι ασφαλίσεις, οι ασφάλειες σε περίπτωση μεγάλων κινδύνων θα έχουν μία ε, αντασφάλιση και θα πληρώνονται ε, τέτοια πριμ, η οποία θα οδηγούνται στην κεφαλική, κεφαλαγορά. Και σε αυτά συγκαταλέγεται και το ίδιο κεφάλαιο. Γι' αυτά χρειαζόμαστε χρόνο και ίδιο κεφάλαιο. Θα ήθελα να μας ε, διευκρινίσετε λίγο Πώς το φαντάζεται αυτό το σύστημα. Λέτε ότι το αμερικανικό μοντέλο ε, ισχύει ήδη. Τι σημαίνει όμως ακριβώς. Και τι γίνεται όταν υπάρχουν ελλείμματα. Ποιος αυθύνεται για τα ελλείμματα αυτά. Ποιος θα διαθέτει το ίδιο κεφάλαιο. Κάτι άλλο μιλήσατε για ε, λύματα, για πλεονάσματα και τέτοιες ε, περιπτώσεις που υπάρχουν πλεονάσματα μπορούμε να πληρώσουμε φυσικά παραπάνω. Αν όμως δημορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, συνάδελφε διακόπτη ο Πρόεδρος. Δύο δευτερόλεπτα θα δούμε ακόμα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα, αν το ευρώ Όπω αναθυνέματα θα έχουμε τερμηνία, λέει ο Πρόεδρο. Πολύ απλά αυτό ισχύει. Πολύ απλά θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονικό όριο. Είχατε το χρόνο που σα αναλογεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όντως, όπως σας είπα, ένα ενιαίο σύστημα ασφάλειας ανέργων στην Ευρώπη δεδομένων των 27 διαφορετικών παραδοσιακών δομών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας δεν είναι κάτι το πολύ πιθανό γιατί είναι διαφορετική και η κατάσταση και θα ήταν δύσκολο να οικοδομηθεί κανένα τέτοιο σύστημα. Ιδιαίτερα επειδή έχουμε καταστάσει σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η ασφάλεια στον μακροπρόθεσμα ανέργων δεν υπάρχει καν. Θα πρέπει καταρχάς να υπάρχει κάτι τέτοιο και να υπήρχε η διανάληψη ευθυνών για τέτοιες περιπτώσεις, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν λίγο πιο επισταμένους ε, τι ισχύει σε ό,τι αφορά τις επιστροφές των πιστώσεων αυτών. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε διάφορες μορφές, γιατί ε, δεν ε, αποκλείεται η περίπτωση μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, όμως λειτουργήσε το σύστημα παρά και τις διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις που επικρατούσαν στις διαφορετικές χώρες. Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ προσωπικά θα σύστηνα να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε τι μπορούμε να διδαχθούμε και νομίζω ότι ένα συνδυασμό των στοιχείων των οποίων ε, ανέφερα θα άξιζε τον κόπο. Προφανώς δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα μιας ε, διαρθρωτικής κρίσης η οποία θα έπλετε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε καλύτερα σε κλειδονισμούς σε μεμονωμένες χώρες και να παρακολουθούμε και χώρες όπου υπήρχε επιτυχία. Εγώ, για παράδειγμα, ως πρώην Υπουργός Εργασίας στην Γερμανία, θεωρούσα ε, πολύ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε περιπτώσεις ύφεση αυξάναμε το επίδομα ανεργίας προκυκλικά. Αυτό σε περίπτωση ενός συστήματος ασφάλισης θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την ε, οικονομική, τον οικονομικό κύκλο. Να έχουμε επίσης υπόψη ότι έχουμε δύο πράγματα τα οποία συνδέονται. Το ευρώ, το κοινωνόμισμα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει κοινωνόμισμα, μόνο υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Thank you. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βολφ Κλίντς. Κύριε Υπουργέ, πριν από κάποιες εβδομάδες βγήκε η Ελλάδα από το τρίτο πρόγραμμα και είχα την ευκαιρία στα πλαίσια μιας ε, αντιπροσωπείας ε, να συνομιλήσω με εκπροσώπους και της κυβέρνησης και της Ελληνικής Βουλής. Και η αρχική αισιοδοξία δυστυχώς εξαφανίστηκε αρκετά γρήγορα. Μου φαίνεται ότι τα έσοδα στο μέλλον θα είναι ε, αρκετά ρεαλιστικοί... σε ό,τι αφορά το πλεόνασμα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και το καθεξής. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και εσείς ε, και ο κύριος Μοσκόβηση μας είπε στο Στρασβούργο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει τέταρτο πακέτο για την ε, υποστήριξη της Ελλάδας, ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πώς ε, θα ψηφίζατε όμως αν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής σας η Ελλάδα χρειαζόταν και ζητούσε βοήθεια, επιπλέον βοήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση της Δανίας και της Βρετανίας δεσμεύτηκαν να εισαγάγουν το ευρώ. 7 απομένουν ακόμα. Με την εξαίρεση της Βουλγαρίας, καμία από τις χώρες αυτές όμως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση. Τι θα κάνετε εσείς και οι συναδελφοί σας για να σπρώξετε αυτά τα κράτη-μέλη που έχουν δεσμευθεί να προσχωρήσουν στο ευρώ σε ό,τι αφορά τρίτον ε, τον ε, φόρο συναλλαγών για τη μαζική, μαζικό περιορισμό των παραγωγών, που φτάνει το εμπόριο τους σε ύψη 3 εκατομμυρίων. Ο γαλλικός φόρος σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται για να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για φόρο επί του κύκλου εργασιών. Πολλές ερωτήσει λοιπόν ακούσαμε. Να απαντήσω εν συντομία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον στόχο, τον φόρο των ε, συναλλαγών κάλιο πέντε και στο χέρι, θα έλεγα, παρά δέκα και καρτέρι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Το δεύτερο, η Ελλάδα βγήκε από το πρόγραμμα, είναι στο σωστό δρόμο. Δεν συμφωνώ με, τη σκεπτικό, με τον σκεπτικό τρόπο για τις δισταγμού που εκφράσατε σε ό,τι αφορά το μέλλον. Πιστεύω ότι κοιτώντα τα πράγματα κατά τη διάρκεια τη κρίση τα τελευταία χρόνια, τα σενάρια ανάπτυξης είναι πιο πιθανά από τα απεσιόδοξα. Αυτά που πέτυχε λοιπόν η Ελλάδα πριν από την κρίση θεωρώ ότι θα φανούσε κάποια χρόνια. Και πιστεύω ότι αυτές οι προπτικές για την Ελλάδα και την ανάπτυξή της δεν είναι στον αέρα. Και νομίζω ότι θα υπάρξει ανάκαμψη στην Ελλάδα. Και αυτό πραγματικά το εμπιστευόμαστε σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. Δεν θεωρώ ότι θα χρειαστούμε περαιτέρω πρόγραμμα. Και να πω ότι είναι μια επανειλημμένη επιτυχία των μηχανισμών σταθεροποίησης τους οποίους έχουμε στην Ευρώπη και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Είδαμε τι ικανότητες έχουμε και αυτό διαφαίνεται εκ νέου. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση, αλλά στα τελική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε το μηχανισμό σταθερότητας, την καλή μας ε, φήμη και το κύρος μας. Και νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή που μπορούν πλέον να λάβουν μόνοι τους να συνεχίσουν. Για την προσέγγιση στην Ευρωζώνη. ρωτήσατε και αυτό. Νομίζω ότι θα πείσουμε από μόνοι μας και θα υπάρξει μία επίδραση του γεγονότος ότι 85% του προϊόντος προκύπτει από την Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες, θα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Ευχαριστούμε, Έρνες Τουρτασούν. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, που είστε σήμερα μαζί μα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κλίντ και θα ρωτήσω και εγώ τι γίνεται με το EFTD. Εάν εξαιρείτε και αυτό από το φόρο, θα είναι ε, λανθασμένη ονομασία το EFTD. Και μετά έχω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Για την ε, ε, αναχώρα υποβολή εκθέσεων, το CCTB. Ε, Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο το παρακολούθησε στενά το θέμα. Στο τελευταίο όμω τριμερή το μπλόκαρε η Γερμανία που δεν ήταν έτοιμη για διαπραγματεύσει. Ξέρω ότι οι Γερμανοί, οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε έχουν το CBCR στο δικό του ε, προεκλογικό ε, και γενικότερα στο πλάνο τους. Ε, ποια είναι η θέση του Υπουργείου σα για το σχέδιο αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε για το CBCR και μετά για ε, το, για το ρόλο του Κοινοβουλίου στο μέλλον για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο διακυβερνητική συνεννόηση χωρίς καμία λογοδοσία από αυτό το σώμα. Νομίζω μια μεγάλη πλειοψηφία εδώ θέλει να υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος για τη μελλοντική λειτουργία του Ταμείου Και θέλω να γνωρίζω εάν μπορούμε να υπολογίζουμε σε εσά ω Υπουργό Οικονομικών, για να έχουμε ένα τέτοιο ταμείο το οποίο να ελέγχεται και από το Κοινοβούλιο και να υπάρχει λογοδοσία. Σα ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το θέμα των εκθέσεων αναχώρα, αυτό λειτουργεί μόνο όταν συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Αυτό αφορά και τις χώρες και τις επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν υπάρχουν εκθέσεις, δεν θα σημειωθεί πρόοδος. Και άρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση η οποία να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Αν καταστρέψουμε τις βάσεις ε, για να παίρνουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν θα πετύχουμε τίποτε. Άρα, να προσέξουμε προκειμένου να είναι αποτελεσματικό το εργαλείο το οποίο θα δημορφωθεί στη τελική ανάλυση. το οποίο θα γίνεται αποδεκτό και από τις χώρες και από τις επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσει παγκόσμια το σύστημα αυτό. Αυτό θα υποστηρίξω, αυτή την προσεκτική οδό, σε ό,τι αφορά τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα και των θεμάτων που συνδέονται με αυτό. Θεωρώ ότι ενδεχομένως συμφωνούμε ότι σε πρώτη ανάλυση θα ήταν δυνατή μία μεταρρύθμιση που θα συνδέεται με το διακυβερνητικό σύστημα υπάρχουν ε, σημαντικές ε, νομικές αμφιβολίες κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λέω ήπια, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Αλλά θα αντιμετωπίσαμε σίγουρα μεγάλες δυσκολίες αν ακολουθούσαμε άλλη οδό στην παρούσα φάση. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η μεταρρύθμιση να γίνει στο υπάρχον πλαίσιο, να γίνει τροποποίηση της συνθήκης και να γίνει διακυβερνητικά η μεταρρύθμιση και σε δεύτερο βήμα να προσπαθήσουμε να μπει αυτό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο βήματα είναι σημαντικά. Αν υπάρχει ένα καλό ESM, ένας καλός και εύρυθμος ε, μηχανισμός σταθερότητας, μια τροποποίηση της συνθήκης δεν θα α, επιφέρει κριτική από κάποιες ε, χώρες, το οποίο συμβαίνει συχνά όταν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τα φορολογικά. Να δούμε λοιπόν το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, φυσικά το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και τι αποτελέσματα θα έχει είναι άλλο θέμα. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε έξυπνα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του καθεστώτος και στη συνέχεια ενδεχομένω να αλλάξει μέσω τροποποίηση της συνθήκης το κοινωτικό δίκαιο. Να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Σε πολλά κράτη-μέλη για τα οποία δεν έχω ευθύνη, αλλά και η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα. Υπάρχουν σημαντικά συνταγματικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν σε ό,τι αφορά το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Γι' αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έγιναν διαβουλεύσεις ε, για το σύστημα μετοχών, το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει ένα θέμα ουσιαστικά. Κατά πόσον αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε άλλο επίπεδο μπορούν να επηρεάζουν ε, την νομοθεσία για την κατάρτιση προπολογισμού των εθνικών κοινοβουλίων και κατά πόσον μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί μιλάμε για αποφάσεις τις οποίες στη τελική ανάλυση μπορούν να πάρουν μόνο οι αιρετοί βουλευτές. Αυτό λοιπόν το θέμα ε, επανειλημμένα ανακύπτει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και από το Γερμανικό Δικαστήριο και από άλλα δικαστήρια άλλων κρατών μελών. Το θέμα λοιπόν του κατά πόσον ε, πλήττεται το δικαίωμα κατάρτιση προπολογισμού από τις εθνικές πουλές. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην το κοιτάξουμε από πλευρά σε της παγκόσμιας οικονομίας, να μην να... Α, ξεπεράσουμε ζητήματα Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτισμού, γιατί εκεί πέρα θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πιο σκόπιμο να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που σας περιέγραψα προηγουμένως. Thank you. Ευχαριστούμε. Είπαμε ξεκάθαρα ότι είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκριθεί, θα στηρίξουμε το υπάρχον πλαίσιο που αναφέρει τον ε, δραστήριο και αποφασιστικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο κύριος Σίρντεβαν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Υπουργό που απαντάει στα ερωτήματα των ε, βουλευτών και έτσι νομίζω αποδεικνύεται ότι η σοσιαλδημοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή και δεν χάνονται όλα στη μάχη μεταξύ Τσέσου και Τσεντεού και Αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερα είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης. Είπατε και παραθέτω ότι ένας ε, Γερμανός Υπουργός Οικονομικός είναι Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Και νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί στην εξή ερώτηση. Ενδεχομένως να συμφωνήσουμε ότι το, ευρωπαϊκό εμπορικό, το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα και ιδιαίτερος... Ναι, μιλάω κάπως γρήγορα. Εντάξει, θα ερεμήσω, θα χαλαρώσω. Σας το υπόσχομαι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδεχομένως να συμφωνήσουμε ότι το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα ε, ξεκινά διαδικασίες κρίσεως στην Ευρωζώνη ιδιαίτερως ε, και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της Γερμανία στις δημόσιες υποδομές ε, και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της ιστορικής αγοράς, επένδυση ε, σε άλλες υποδομές για να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα και στον ε, στρατιωτικό τομέα η γερμανική κυβέρνηση Δεν μπορεί δηλαδή η απάντησή σας να είναι ε, ένα στατιστικές επενδύσεις για το μέλλον. Επίση, κάποιοι θα λέγανε ότι συνεχίσετε την πολιτική λιτότητα στο Σόιμπλε. Πριν ε, λέγατε ότι δεν έχουμε χρήματα. Τώρα σα λέω ότι ε, μα ναι, υπάρχουν χρήματα. Εκατοντάδε ε, δισεκατομμύρια τα οποία ε, φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να τα μαζέψουμε αυτά τα χρήματα. Άρα, τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον εδώ, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα του υψηλού κατατατού συντελεστέ φορολόγηση των εταιριών. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει τουλάχιστον. Να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, το θέμα της ε, πολιτικής ε, κατάρτισης του προπολογισμού και τι επενδύεται. Να σας πω ότι ο γερμανικός ε, προπολογισμό είναι πολύ επεκτατικός ε, και το τρέχον έτος και στις επόμενα χρόνια σε σχέση με το 2017 και το σχέδιο του 2018 που καταρρίστηκε ο προπολογισμό το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την επόμενη νόμισμη, την επόμενη περίοδο έχουμε επιπλέον 50 δισεκατομμύρια ε, δαπάνες, το οποίο είναι δυνατόν με περισσότερα έσοδα. Δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό που θα αναμενόταν την χρήση των παραπάνω εσόδων για τη μείωση των ελλημάτων και συνεχίζουμε να κάνουμε υψηλές επενδύσεις. Και οι μεγάλες αυξήσεις που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια θα παραμείνουν σε τέτοια επίπεδα ε, πρόσθετα δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια σε σχέση με τους προπολογισμού των, των τελευταίων χρόνων και υπάρχει η δυνατότητα και περαιτέρω αύξησης και για την ε, κοινωνική συνεργασία, για τη φύλαξη παιδιών, πολύ ψηλές δαπάνες για τους πολίτες για μείωση των ε, κοινωνικών εισφορών, για σταθεροποίηση των συντάξεων και για τους επιπλέον φόρους. Εξασφαλίσαμε ότι θα έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συμβάλλουμε σε συνέχιση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τα ξέρετε, μεγάλο τμήμα των δημόσιων υποδομών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι είναι σωστό, αλλά νομίζω ότι καλά θα κάναμε να το λέμε και όλα ανοιχτά, γιατί κάποιοι ασκούν κριτική ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να το διευκρινίζουμε αυτό και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για το μέλλον σε ό,τι αφορά την αύξηση των μισθών. Έχει δρομολογηθεί και ένα σημαντικό ποσό της αύξησης των ε, φοροεσόδων έχει να κάνει με την αύξηση των μισθών. Ό,τι σημαίνει αυτό και με την ανάπτυξη. Το πακέτο λοιπόν που περάσαμε και την απελευθέρωση πόρων από το πακέτο αλληλεγγύης από την Γερμανική Επανένωση. Αυτά για να τονώσουν την κατανάλωση και πιστεύω ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Σα ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά την εξηγήση των τραπεζών. Αν κατάλαβα σωστά, προβλέπετε το ESM στο μέλλον να χρησιμοποιείται ε, μόνο ω ε, τελική λύση. Το ESM είναι ένα ε, θέμα το οποίο διακυβεύεται σε ό,τι αφορά την λειτουργία του νομισματικού ταμείου. Μία τελική λοιπόν τέτοια εγγύηση για τις τράπεζες μέσω του, τραπεζικού μηχανισμού θα ήταν μέσω του μηχανισμού ντόμινο, όπως και με την Ελλάδα. Και μιλάμε λοιπόν για μια συστημική τραπεζική κρίση, αλλά το ESM είναι πάρα πολύ μικρό για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Ακόμα και η εξυγίανση η Γερμανική Τράπεζα, για παράδειγμα, κόστισε 14 δισεκατομμύρια και πλέον. Το ESM λοιπόν δεν αρκεί για την επίλυση τέτοια συστημική κρίση όλη τη Ευρωζώνη και ακριβώ επειδή υπάρχουν αυτά τα όρια, έχουμε και μία γραμμή διάσωση στην ΕΚΤ. Euro System Resolution Liquidity. Αυτό αποφασίστηκε λοιπόν και στην. Ε, ναι, ναι, ναι, τα λέω γρήγορα. Θα διαβάζω γρήγορα. Να προσπαθήσω και λίγο πιο αργά. Το Resolution Landing Facility της ε, Bank of England. Η ερώτηση λοιπόν που έχω να σας απευθύνω. Η τραπεζική διάσωση στα μάτια της γερμανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί μόνο δημοσιονομική λειτουργία και η λειτουργία διάσωσης της ΕΚΤ δεν είναι αντίθετη με την εντολή της ΕΚΤ απάντηση. Τα τελευταία χρόνια κάναμε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Νομίζω λοιπόν ότι αν αντιληφθούμε όλα τα βήματα τα οποία έχουν γίνει από το 2008 έχουμε προχωρήσει πολύ. Γιατί υπήρχε συστημικός κίνδυνος Και αυτά που έκαναν οι Αμερικανικέ τράπεζε και το Αμερικανικό σύστημα δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε στην Ευρώπη. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν πολλά εργαλεία. Και αυτό αποτελεί πρόοδο. Μεταξύ των εργαλείων αυτών λοιπόν τον ε, μηχανισμό εξυγίανση τραπεζών, για παράδειγμα, ο οποίος αναπτύχθηκε, που μπορεί να συμβάλλει στις τράπεζες που έχουν συστημική σημασία και στην τελική ανάλυση θα είναι τα παπτικά όργανα αυτού του μηχανισμού κατά πόσον πρόκειται για συστημική κρίση για τις τράπεζες και κατά πόσον υπάρχουν συνέπειες για όλη την ε, Ένωση και έχει επίσης και ιδιαίους πόρους 8% που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους πιστωτές ε, και για μια κάποια αναδιάρθρωση των τραπεζών. Για να δούμε κατά πόσον μήπως ε, πέρα από την εξυγίανση των τραπεζών μπορούμε να αποφύγουμε και συστημικούς κινδύνους. Δεν υπάρχουν αλγόριθμοι, είναι αποφάσεις που λαμβάνονται για το τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση και η απάντηση μπορεί να είναι αρνητική ή θετική. Και πέραν αυτού υπάρχει και μία τελευταία εγγύηση σε ό,τι αφορά την ικανότητα εξυγίανσης του μηχανισμού αυτού. όπου το εξεταζόμενο στοιχείο δεν είναι η ικανότητα δανεισμού του ESM, αλλά η ικανότητα του μηχανισμού εξυγίανσης. Ένα μετρήσιμο μέγεθος. σε ό,τι αφορά την δυνατότητα άμεση επανακεφαλαιοποίηση από το ESM. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε γιατί δεν μπορούσε έτσι και αλλιώ να εφαρμοστεί. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ σταθερό και το οποίο θα μπορέσει να αντιδράσει με αποτελεσματικό τρόπο. Γιατί υπάρχει εκεί και διακυβέρνηση. Θα πρέπει γρήγορα να αποφασίζονται τέτοια στοιχεία, να λαμβάνονται αποφάσει. Καθιερώνται λοιπόν αυτές ε, οι δυνατότητες, αλλά όλα αυτά θα αποφασίζονται κατά περίπτωση. Δεν θα υπάρχει κάποια νομική πρόβλεψη. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποφασιστούν. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για ρευστότητα, μπορούμε από συστημική ε, άποψη, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει στην ε, επόμενη περίοδο. Θα πρέπει να συζητήσουμε πιο πολύ τα θέματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτά είναι τα πλέον κατάλληλα. Thank Κυρία Κάπελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας. Χθες είχαμε τον πρόεδρο του, της Αυστριακής Προεδρίας, του ΙΚΟΦΗΝ, ο οποίος μας δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να δούμε την αρχή και τον οδικό χάρτη για το μείωση του κινδύνου και τον επιρρυθμό του κινδύνου. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό πακέτο, σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλα βήματα στα πλαίσια του backstop στο SRF. Συγκεκριμένα και σημαντικά στοιχεία είχαμε και τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος μας είπε ότι στο θέμα μείωση του κινδύνου έχουν λεφθεί ε, και έχουν ε, υλοποιηθεί πολλά μέτρα τα οποία προωθούν την ελεγγύη. Άρα από πλευρά σας ακολουθείτε την άποψη του Συμβουλίου ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τη μείωση και μετά τον περιορισμό, τον του κινδύνου. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον ε, φόρο συναλλαγών, η Αυστρία τα τελευταία χρόνια Η Αυστρία κοιτάει το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ εμπισταμένο. Και ακούσαμε ότι θα ήταν πιο σωστό να ακολουθηθεί μια καθολική λύση παρά μια μικρή, μικρής κλίμακας λύση. Εσείς μιλάτε τώρα για το γαλλικό μοντέλο. Θα κάνετε συγκεκριμένα βήματα για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και κατά πόσον θα ακολουθηθεί το γαλλικό μοντέλο. Τρίτη ερώτηση είπατε ότι θα είναι απαραίτητο να υπάρχουν νέε δημοσιονομικές ικανότητες για τη σταθεροποίηση. Το InvestEU πιστεύετε ότι είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ενταχθεί στο Πουδουπού. 650 εκατομμύρια ευρώ έχει προοικοδότηση. Είναι αυτό ένα μέτρο λοιπόν για τις νέες δημοσιονομικές ικανότητες. Η απάντηση. Νομίζω ότι η μείωση του κινδύνου και η αλληλεγγύη είναι δύο στοιχεία που πάνε χέρι-χέρι. Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι όλοι κατανοούμε ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε αλληλοκατηγορώντα Δεν συμβαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο γιατί οι μεν λένε μείωση του κινδύνου και οι άλλοι λένε επιμερισμός του κινδύνου. Γιατί αυτό πολύ απλά διαιωνίζει το πρόβλημα. Θα ήταν μια καλή πρόοδο να πούμε ότι όλα είναι σημαντικά και χωρί τη μείωση του κινδύνου το τραπεζικό πακέτο δεν πρόκειται να αποδώσει καρπούς και αυτό συνδέεται και με τη μεταξέλιξη του ESM. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά αντίφαση μεταξύ των δύο στοιχείων. Αν ε, φυσικά επιθυμούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα, πρέπει να κάνουμε και τα δύο μαζί. Και τότε θα λειτουργήσει το σύστημα. Άρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι να σταματήσουμε να μιλάμε και να ακολουθήσουν πράξεις σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου. Θα πρέπει να πετύχουμε και άλλα πράγματα παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί πρώτοι Να δρομολογηθούν λοιπόν όλα αυτά. Φόρος συναλλαγών. Να δούμε. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ακολουθούμε μία χήμερα. Να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε συγκεκριμένα. Μπορούν να λειτουργήσουν λοιπόν αυτά εάν τα συνδέσουμε με τη συζήτηση και το θέμα του προπολογισμού. Τότε θα έχουμε επιπλέον δυνατότητε σε ό,τι αφορά τι συγκεκριμένε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που ακολουθούν τον γενικότερο στόχο, αλλά δεν έχουμε ακόμα την πρόταση σε τελική ανάλυση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα ομαδοποιώντα ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις λίγο. Η Έστερ Ντελάγκε έχει το λόγο. Για το ίδιο, κυρία Υπουργέ, ήσασταν α, λίγο μυστήριος θα έλεγα. Αναφερθήκατε στον οδικό χάρτη που περνά από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις και είπατε ότι συνδέεται και ότι εδώ σε αυτό το σώμα υπάρχουν πολλές απόψεις σε σχέση με την δομή και τον χρονισμό του Ίντις, αλλά μια μεγάλη πλειοψηφία εδώ πιστεύει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Οπότε λοιπόν ποια είναι αυτά τα θέματα στα οποία λίγο αναφερθήκατε, να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος και δεν πιστεύετε ότι με τη σωστή αιρεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις θα μπορέσει το ίντις να παράσχει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απαιτείται και να επιτρέψει επίσης Ε, τώρα για το δεύτερο θέμα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει ένα βάρος, ένα ιστορία όπως είπατε εσείς. Έχουμε να κάνουμε με χώρες οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε το παρελθόν κάθε χώρας ξεχωριστά. Φάιτσέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη χαρά μου που σας συναντώ και θα ήθελα να ξεκινήσω με μία παρατήρηση. Πολλοί είναι συνάδελφοι ε, συμφωνούν σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε με τα θέματα της αντασφάλισης. Πώς μπορεί να οργανωθεί όμως αυτή η δραστηριότητα στον 21ο αιώνα υπάρχουν θέματα τα οποία εκκρεμούν και άπτονται ας πούμε της μετανάστευσης ε, του εξωτερικού ελέγχου των συνόρων, του ελέγχου μάλλον των εξωτερικών συνόρων, της άμυνας. Πώς θα μπορέσετε να τα συνδυάσετε όλα αυτά έτσι ώστε στην παρούσα συγκυρία της ΚΕΠΑ και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων Μήπως θα υπάρξουν διαφορετικές πορείες από τα κράτη-μέλη, γιατί είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν όλα ε, την ίδια πορεία. Σκύρτσος. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό για το επίπεδο της επιχειρηματολογίας του και για την ευρωπαϊκή του προσέγγιση. Ε, Θέλω όμως να του θέσω ένα θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος, γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ήταν να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα, στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος και γι' αυτό είχε προτείνει πολύ σκληρά μέτρα. Τελικά έφυγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος, αλλά μείνανε τα μέτρα που πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα για το πολιτικό σύστημα. Είναι για παράδειγμα σαν να λέει ο υπουργό εκεί που εκλέγεται ότι πηγαίνει καλύτερα η οικονομία στο Αμβούργο ή στη Γερμανία, ε, αλλά από 1η Ιανουαρίου θα μειωθούν 14% κατά μέσον όρο οι συντάξει. Αυτό δεν γίνεται στην πολιτική, δηλαδή δεν γίνεται να περιγράψει μια κατάσταση και να πηγαίνει προ την αντίθετη κατεύθυνση. Επομένω, έχουμε πολύ σκληρά μέτρα τα οποία μπορεί να βγαίνουν σε επίπεδο οικονομικών εκτιμήσεων, αλλά κατά την άποψή μου δεν βγαίνουν σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής διαχείρισης. Είναι δύσκολο για τη σημερινή κυβέρνηση, εμείς είμαστε στην αντιπολίτευση, μπορεί να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, αλλά θα είναι εξίσου δύσκολο και για μας. Άρα θέλουμε από το Eurogroup περισσότερη κατανόηση και πιο ελαστική προσέγγιση στα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα. Μπορεί να βοηθήσει ο υπουργό προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για τι διάφορε αυτέ ερωτήσει. Να προσπαθήσω να απαντήσω. Όταν συζητάμε το ΕΔΙΣ, ένα πράγμα θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά. έχουμε ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Ε, αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι τράπεζες περνούν από ένα ευρωπαϊκό σύστημα υποπτίας σε ό,τι αφορά την εξυγίανση. Το θέμα είναι τι θα γίνει πριν και μετά, σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Λίγο πολύ υλοποιείται και εφαρμόζονται σωστά αυτός ο κύκλος. Όταν θα υπάρξει το έντις, θα υπάρξει διακυβέρνηση από τα κράτη-μέλη σε πρώτη φάση. Και εδώ υπάρχει μία διαφορά. Δεν θα παίρνει απόφαση ένα θεσμικό όργανο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών. Πάντα θα έχει ευθύνη χωρίς να αποφασίζει κάποιος. Και οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίζουμε θα είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Γιατί θα προσθεθούν και οι κίνδυνοι τις οποίες δεν γνωρίζουμε καν σε ό,τι αφορά τις τεχνικές αλλαγές. Θα μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα κάπου, να λειτουργήσει ως τράπεζα, να χρησιμοποιεί μέσα fintech σε όλη την Ευρώπη και αυτό θα έχει κίνδυνο. Κινδύνους μάλιστα που θα ξεπερνούν ακόμα και αυτά που μπορούμε να φανταστούμε στην παρούσα φάση. Πώς ε, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κοινούς κανόνες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το έντι, Θα πρέπει να συζητήσουμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις πρακτικές καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος, να κοιτάξουμε το θέμα των κρατικών ομολόγων, και τις τραπεζικούς ισολογισμούς. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να επιληθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα βάλουμε στην ατζέντα. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και χαίρομαι που δηλώνουμε ότι θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δεν είναι όμως απλά και ξεκάθαρα και η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στο μηχανισμό εξυγίασης των τραπεζών έχουμε ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που δεν την έχουμε στο ΕΝΤΙΣ. Έχουμε εθνικές, εθνικά συστήματα διακυβέρνησης με εντελώ διαφορετικούς όρους. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα τώρα. Θα πρέπει στόχος μας να είναι η μείωση τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα στόχο ο οποίος θα αποτελέσει και την κατεύθυνσή μας και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και σε ιστορικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι εποπτικές ε, δομές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τις τραπεζικές αρχές επί κάποιων κατευθυντηρίων γραμμών. Ο μηχανισμός εξυγίανσης των τραπεζών και το έντις θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε καλές νομικές συνθήκες προκειμένου οι πιστωτές μπορούν να αγοράσουν ε, θέσεις και να συμμετέχουν ε, γιατί Μία τράπεζα η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιστροφή των ε, καταθέσεων θα αποτύχει γιατί απλά δεν υπάρχει η εγγύηση αυτή και πολύ, κανένας, πολύ απλά κανείς δεν της δίνει χρήματα. Και εδώ τα νομικά καθεστώτα σε κάποιες χώρες απέχουν από αυτό που θα θέλαμε και από αυτό που θα περιμέναμε. Βλέπουμε λοιπόν τα ποσοστά σε ό,τι αφορά την πώληση τέτοιων πακέτων χρεών και όταν βλέπουμε 10% αυτό σημαίνει ότι το σύστημα τη χώρα, το τραπεζικό σύστημα, το σύστημα δικαιοσύνη δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε τέτοιε περιπτώσει και θα πρέπει να κάνουν την, τα μαθήματά του οι χώρε αυτέ. Το θέμα τώρα των ε, ευρωπαϊκών αξιών και του πολιτισμού δημοσιονομικών ε, προπτικών. αν μείνουμε στο 1% του κοινωνικού προϊόντος, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία που θα σημαίνει μεγάλη αύξηση σε πολλά κράτη και ξέρω ότι αυτό έχει να κάνει με τις μεγαλύτερες γραμμές προπολογισμού των εθνικών δαπανών και γι' αυτό ελπίζω ότι οι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν ε, μια καλή ισορροπία για να μην προωθήσουν το λαϊκισμό σε κάποιες χώρες. Αλλά για το πλαίσιο αυτό έχουμε κάποιο περιθώριο σε ό,τι αφορά την πολιτική, την εξωτερική, τη μετανάστευση, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της έρευνας και της κοινωνίας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν βασική σημασία. Έχουν ρόλο κλειδί και θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και στο μέλλον. Πολύ μεγαλύτερο από ότι και σήμερα. Για την Ελλάδα η ερώτηση. Και ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι κάνουμε. Συνοδεύουμε την επιστροφή της Ελλάδας στις οικονομικές αγορές. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Αυτό το βήμα εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνη, οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Αν δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη, ούτε οι πολίτε ούτε οι επιχειρήσει, ούτε η διεθνή αγορά, ούτε τα άλλα κράτη, η επιστροφή στι αγορέ θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό οι συμφωνίε που έχουν ληφθεί, που έχουν γίνει να τηρηθούν στην εκτέλεση του προγράμματο, ανεξάρτητα από το ποιο είναι στην κυβέρνηση στην, στην Ελλάδα. Γιατί οτιδήποτε άλλο πιστεύω ότι δεν θα λειτουργούσε. Και γι' αυτό λοιπόν. Δεν έχουμε εμπειρίε, αλλά α μην το δοκιμάσουμε, γιατί μπορεί να είναι πολύ μεγάλο το τίμημα. Να υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την επανακεφαλοποίηση του ESF κτλ. να προχωρήσει κομμάτι, κομμάτι για την ανάλεψη πιστώσεων στις αγορές και για να υπάρξει η ανάπτυξη. Και ένα καλό καθεστώς είναι η προϋπόθεση. Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να αλλάξουν κομμάτια του προγράμματος που έχει οριστεί. Ότι θα έχουμε νέο περιθώριο ελιγμού με το που βγαίνουμε από το πρόγραμμα, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά θα πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί για να λειτουργήσει το σύστημα. Και εδώ εντάσσεται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει ακόμα ε, πίστοση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Thank you, Pedro Silva Ευχαριστούμε κύριο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, και εγώ σας καλωσορίζω, Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Κυρίως, καλωσορίζω την στήριξή σας στον προπολογισμό, έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης για σκοπό σταθεροποίησης και σύγκλησης. Τρεις ερωτήσεις έχω για τη μεταμόρφωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις είπατε ότι χρειάζεται ένα μεγάλο βήμα με αλλαγές στις συνθήκες. Στις απαντήσεις σας όμως, στα πλαίσια των δηλώσεων και άλλων πολιτικών εθνώντων, είπατε ότι πρέπει να υπάρξουν δύο βήματα. Πρώτα, η αλλαγή στις διακυβερνητικές συνθήκες και μετά σε κατοπινό στάδιο η ενσωμάτωση του μηχανισμού σταθερότητας ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτή η μεταρρύθμιση που θέλουμε να έχουμε για περισσότερο ενωμένη και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μήπως μια μεταρρύθμιση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κανένα δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. τουλάχιστον από αυτό το κοινοβούλιο. Και έπειτα, πόσο μεγάλο είναι αυτό το βήμα, το άλμα που προτείνεται να γίνει, διότι σε μια δεύτερη φάση, βάσει των ε, δηλώσεων Βάσει των δηλώσεων μέσα θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισής του, της governance, στην μεταστροπή του μηχανισμού σταθερότητας σε νομισματικό ταμείο. Τι εννοεί το management εδώ, το governance. Και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου να αξιολογείται η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών χωρίς όμως να ε, παίρνει κάτι από το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε την κατάσταση σε ορισμένα κρατημέλη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι περιθώριο μένει για μια νέα αξιολόγηση, για περισσότερες εκτιμήσεις από ένα νέο χρηματοπιστωτικό ρυθμό. Ευχαριστούμε, ο κύριος Λάγκερ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, επιτρέψτε μου να σας κάνω ένα κομπλιμέντο ως χριστιανδημοκράτης. Ε, τόσα χρόνια δεν ε, έχω δει άλλο υπουργό που να έχει κάνει τόσο γρήγορα και τόσο καλή εισαγωγή στο θέμα του και στο χαρτοφυλάκιο του. Τρεις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την συνασπισμό. Το ESM καταρχά. είπατε ότι θέλουμε να μεταφερθεί αυτό σε κοινωτική νομοθεσία, αλλά στην ε, συμφωνία του συνασπισμού αναφέρεται ότι τα δικαιώματα αυτά θα παραμείνουν ε, απαράλλακτα. Πώ θα τετραγωνίσετε τον κύκλο. Δεύτερον, μιλήσαμε για το φόρο συναλλαγών, ε, έκθεση αναχώρα, όχι για την απαραίτητη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Στη Γερμανία τι γίνεται. Βλέπουμε ότι έχουμε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη ε, για απάτη σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ και οι προτεγραφές BEPS δεν ισχύουν σε ό,τι αφορά τα μικρά κράτη-μέλη. Ουσιαστικά κάνουν φορολογική πολιτική κατά των μεγάλων. Πώς ε, υπάρχουν, τι ευκαιρίες υπάρχουν να αλλάξει αυτά τα επόμενα χρόνια και τι θα πρέπει να πούμε σε ό,τι αφορά και την φορολογική αντίδραση και αλλαγή του Τραμπ. Τελευταία ερώτηση ο ευρωπαϊκό προπολογισμό μετά τον Brexit θα πρέπει να γίνουν αλλαγέ. Έκανε προτάσει ο κ. Σότιγκερ, επικρίθηκαν στη Γερμανία. Πού πιστεύετε ότι διαμορφώνεται η γραμμή στο 1,24% το ανώτατο όριο ή κοντά στο 1,0% βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε, Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον κύριο Σόλτς και εγώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς για τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεστε ε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας για να τροφοδοπτήσουμε σταθεροποιητικά την οικονομία. Για το έμπις. Θα ήθελα να συμμεριστώ μέσα ε, το ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι ευρωπαϊκά όργανα βέβαια ρυθμίζουν ε, τον τραπεζικό τομέα, εποπτεύουν του τραπεζικού τομέα και βοηθούν να λυθούν τα θέματα του τραπεζικού τομέα ενώ υπεύθυνοι για την σωστή εποπτεία, την σωστή ή λανθασμένη εποπτεία, πάντα είναι εθνικά όργανα σε μία πρώτη φάση. Τίθεται το θέμα λοιπόν εδώ του ηθικού κινδύνου και το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν λαμβάνουν και την υποχρέωση να δεχθούν την ευθύνη των για τις αποφάσεις τους αυτές. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί προβλήματα. Ναι μεν θα πρέπει να προχωρήσουμε συνολικά στον τραπεζικό τομέα, καλύτερα ίσως από ό,τι σήμερα, και έχουν γίνει κάποια βήματα, γιατί η κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα, μακροπρόθεσμα δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να διατηρηθεί. Και τώρα σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να εντάξουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια της συζήτησης για το ΕΒΙΣ. Ή θα πρέπει να συνδέσουμε τη συζήτηση για το δημόσιο χρέος με τη συνολικότερη συζήτηση ή θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε με κάποιο τρόπο διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ. οι συνάδελφοι ε, δεν, ε, που ήταν στο Catch the δεν είναι εδώ τώρα. Γενικά χτες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με τα λεγόμενα backstop. Αυτό το οποίο χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι ένα τέτοιο backstop για να είναι αποτελεσματικό εφόσον τα χρήματα τα οποία είναι στο αρμόδιο ταμείο δεν επαρκούν, πρέπει να υπάρχει σωστή εποπτεία. Και δεν θα πρέπει κατά περίπτωση κάθε φορά το Κοινοβούλιο να υιοθετεί μία απόφαση έτσι ώστε να καλυφθούν κατά 100% οι ανάγκες. Πρέπει τα χρήματα να είναι ε, δεδομένα, να είναι διαθέσιμα. Οπότε πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα της διακυβέρνησης και της ε, λήψης αποφάσεων για την ενεργοποίηση του Μπάξοφ. Κύριος Μαριάς. I question in Greek, Mr. Minister. Do translation? Thank you. Κύριε Υπουργέ, η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία τηρεί τις δεσμεύσεις της. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας ρωτήσω επειδή το, ε, στις 14 Μαρτίου του 1942 υπευλήθη ένα αναγκαστικό κατοχικό δάνειο από τις γερμανικές αρχές κατοχής στην Ελλάδα. Ένα δάνειο το οποίο άρχισε να εξοφλεί η Γερμανία με εννέα δόσεις το 1943 και μετά σταμάτησε να το εξοφλεί. Το ερώτημά μου είναι, εσείς ως Υπουργός Οικονομικών, πότε προβλέπετε να συνεχίσετε την εξόφληση αυτού του δανείου το οποίο ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Έχετε προδιαγράψει το στόχο της εξόφλησης αυτής και για πότε προβλέπετε αυτή την εξόφληση του αναγκαστικού κατοχικού δανείου που υπευλήθη το 1942, εξοφλείται με δόσεις το 1943, αλλά είναι ανεξόφλητο ακόμα. Okay. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα αυτά. σε ό,τι αφορά το ESM. Πολλές ερωτήσαμε, ερωτήσεις ακούσαμε για το πώς θα διαμορφωθεί η διακυβέρνηση. Αυτό να το συζητήσουμε. Εγώ να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε επιλογή. να δημιουργήσουμε μια δομή διακυβέρνηση η οποία θα συνδέεται με τα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά τους ε, αποσπασμένους και που συμμετέχουν στο όργανο αυτό. Ό,τι υπόλοιπο, ό,τι άλλο δεν θα εκπληρώνει τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Και γι' αυτό λοιπόν να μην να υλοποιήσουμε, να μην προτείνουμε μια ιδέα η οποία δεν θα είναι υλοποιήσιμη, γιατί υπάρχουν συνταγματικά κολλήματα και έχουν και θέματα σε ό,τι αφορά ε, το δικαστικό του σύστημα και δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην απόφαση ε, των βουλευτών για τον προπολογισμό. Άρα δεν έχει νόημα να κάνουμε καν την απόπειρα να το ξεφορτωθούμε αυτό το στοιχείο. Γιατί για πολλά κράτη-μέλη και για το δικό μου δεν υπάρχει δυνατότητα να ανατεθεί σε άλλον η λήψη απόφασης αυτής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε γρήγορους μηχανισμούς και αποτελεσματικούς ε, μηχανισμούς ε, που θα επιτρέψουν λήψη αποφάσεων σε μία νύχτα, σε ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ήταν λάθος να ελπίζουμε καν ότι θα μπορέσουμε να το παρακάμψουμε αυτό ακόμα και αν προσωπικά το επιθυμούσαμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω εκ νέου έκκληση. Αυτό δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε στον δρόμο. Μόνο λοιπόν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεύτερο θέμα. Το πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε και να κινηθούμε από το Α μέχρι το Β. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν θα ήταν στα πλαίσια του τρέχοντος ε, συστήματος μια συνθήκη των ευρωπαϊκών συνθήκων όπου το ESM θα συμπεριληφθεί όπως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο δηλαδή από τις Ευρωπαϊκές ε, Βουλές θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η σύνθεση. Είναι σημαντική για πολλές χώρες που έχουν την συνταγματική αυτή διάταξη, τον συνταγματικό αυτό περιορισμό. Και δεν υπάρχει δυνατότητα ελεγμού. Αυτά τα δύο βήματα τα οποία συνάπτουν και με τον συνασπισμό και τι συμφωνίε που έχουν ληφθεί στα πλαίσια του συνασπισμού στη Γερμανία. Για τη μεταρρύθμιση τώρα του ΦΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο εδώ. Έχουμε κάποιες προτάσεις ε, που έχουν αναβληθεί, μικρές ε, μεταρρυθμίσει για τη μείωση της ε, φοροαπάτης στο ΦΠΑ. Ελπίζω όλα τα μπλοκαρίσματα τα οποία έχουν προκληθεί και που δεν έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση, έχουν να κάνουν με την ε, ισχυρογνωμοσύνη του καθενός να ξεπεραστούν. Διάφοροι ρώτησαν τι γίνεται με τα κέρδη και τους φόρους. Το BEPS εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ να πω το εξής, ότι αν κοιτάξουμε το αμερικανικό σύστημα φορολόγησης υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και της μετατόπισης ε, κερδών που εν μέρη παραβιάζουν και διεθνείς συμβάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας σε ό,τι αφορά την αυστηρότητά τους και στα πλαίσια του G7 και του ΩΣΑ. λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ε, συμφωνίες που θα ε, επέτρεπαν την διαμόρφωση τέτοιων καθεστώτων. Με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ότι σήμερα. Οι σφορές, επίσης, ε, ε, ακούσαμε και μια ερώτηση για τις σφορές και πόσο υψηλές θα ήταν. Να το θίξω εκ νέου το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι αν κοιτάξουμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι και 1% του κοινωνικού προϊόντος ε, θα σήμαινε αύξηση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και μάλιστα σημαντική αύξηση. Και θα ήταν θεωρητικό. Ακόμα και με το μέτρο αυτό να δούμε τι θα σήμαινε η αύξηση αυτή της χώρες, γιατί μιλάμε για ε, μεγέθη τα οποία δύσκολα εξηγούνται σε διάφορες χώρες. Να μην έχουμε λοιπόν υπερβολικές απαιτήσει και υπερβολικά όνειρα. Είναι σημαντική η διαδικασία αυτή και θεωρώ ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε σχέση και με τους εθνικούς προπολογισμού. Το έντις αυτό ε, θίξατε εκ νέου. Σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε είναι θετικό το ότι το συζητάμε. Συζητάμε δηλαδή το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον, αλλά είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι κρεμή και δεν είναι εύκολο να τα επιλύσουμε. Τα ανέφερα και να σας αναφέρω και ένα περιστατικό όταν ήμουν στην Γερμανικό Κοινοβούλιο και αντιμετωπίσαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την Ισλανδία και το Ισλανδικό τραπεζικό σύστημα, πολλοί πολίτες ε, βγήκαν και είπαν ότι είχαν καταθέσεις στι Ισλανδικέ τράπεζες, τι οποίες και ήθελαν να επιστραφούν. Και είπα ότι κοιτάξτε, δεν έχω ούτε αρμοδιότητε ούτε μέσα, ούτε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα να σας φέρω τα χρήματά σας. Και είχαν κάνει επενδύσεις ε, σε μια χώρα όπου δεν υπήρχε σύστημα ασφάλιση των καταθέσεων με απόδοση 0,5%. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει ότι δεν είναι μηδαμινή σημασία στο κατά πόσον υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε ό,τι αφορά όλα τα ζητήματα τα οποία θίξαμε, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί παντού και η ευθύνη υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια. Είναι πραγματικά πρόβλημα, εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ανάληψης ευθυνών. Τα κρατικά χρέη επίσης αναφέρθηκαν στο σύγκειμενο αυτό και το ανέφερα σε ό,τι αφορά το μερίδιο των κρατικών χρεών στο τραπεζικό ισολογισμό. Το συζητήσαμε αυτό. Αυτό θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Θα μπει στην ατζέντα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω από αυτό. Για την ερώτηση της διακυβέρνησης ε, έκανα συνοπτικά την απάντησή μου και σας παρουσίασα την άποψή μου. Δεν έχω κάτι καινούργιο να πω για το θέμα αυτό. What about my question, Mr. No, Minister? Sorry, sorry. You... What about my question about Mr. the Mr. Marias. German loan? Thank you very much. So, would like to thank very... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Υπουργέ Σόλτς. και για τα τόσο περίπλοκα θέματα που καλύψατε. Σας ευχαριστούμε για τη φιλευρωπαϊκή σας στάση και ευχαριστούμε και για τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το διάλογο και να τον συνεχίσουμε με το Συμβούλιο. Όπω σα ενημερώσαμε στην αρχή τη συνεδρίαση, λόγω τη ε, κινητοποίηση των διερμηνέων θα σταματήσει η διερμηνία στην προβλεπόμενη ώρα που ήταν 12 για αυτή τη συνεδρίαση. State with the appropriate parliamentary control by, by national parliaments. That's why when we took a public position, we said that when we integrate in the union law, we support the EIB model. So we don't want to take the place of national parliament because we know that these are money that come from the national budget. So on this we are crystal clear.